Okay, Συνάλφοι, να ξεκινήσουμε. Από τις 9 το πρωί έχουμε αρχίσει και όσοι ήταν συντονιστές. Είδαμε και τον, τους υπουργούς ε, στο διάλειμμα. Λοιπόν, σημείο 21, παρουσίαση ε, ο, ο, ΣΑΝΤΑΚ, μια αξιολόγηση ομοτήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε ότι είχαμε κάποιους ερευνητές που είχαν στην Επιτροπή μας από τον ΩΣΑ την περασμένη φορά και άκουσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρουμε και εμείς δηλαδή στην αξιολόγηση ομοτήμων είναι μια αξιολόγηση ομοτήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε για την πολιτική ε, για το 2018 την πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη φαντάζομαι ότι έχετε λάβει σχετική πρακτικά αντίγραφα της έκθεσης εγκρίθηκε το φθινόπωρο, δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο. Είχαμε και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν καλό ε, να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση ομοτήμων, διότι, διότι είμαστε στη φάση της έγκρισης του νέου πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη. Έχουμε πολλά να μάθουμε από το παρελθόν τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά και πρέπει να διορθωθεί. Να αντλήσουμε λοιπόν κάποια διδάγματα από αυτή τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την όσα, τον όσα. Είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που βρίσκεται εδώ η ΩΣΑ. Χαίρομαι που είναι μάλιστα εδώ ένα πρώην συνάδελφο, πρώην Ευρωβουλευτή, ο Ζόρζε ο Ζορζ Μορέιρα Ντασίλβα, υπεύθυνο ε, για τα ζητήματα συνεργασία στην ανάπτυξη στον ΟΣΑ ήταν ευρωβουλευτή ε, στο ΕΛΚ, για το ΕΛΚ μάλλον, από το 1999 στο 2003 πριν αναλάβει κυβερνητική θέση στην Πορτογαλία. Έχει λοιπόν μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την πολιτική ανάπτυξη, ε, αλλά και την περιβαλλοντική πολιτική. Ήταν ε, υπεύθυνο στη χώρα του. Έχει εργαστεί και για τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Είναι εδώ και ο Κάρο, Μιαμότο που εργάζεται στην ίδια διεύθυνση του ΟΣΑ για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Στη συνέχεια θα μιλήσει η Κόνκορτ ε, και βεβαίως στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που μου δίνετε την δυνατότητα να παρουσιάσω την αξιολόγηση ομοτύπων, ομοτήμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του DAC, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Πριν από 54 χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή, είναι πλέον θεσμός. Ε, η αξιολόγηση ομοτήμων ε, είναι κάτι από τον οποίο όλοι έχουμε να μάθουμε, από την εμπειρία αυτή. Να σας πω επίσης ότι αυτή η αξιολόγηση ομοτήμων έχει αντίκτυπο. 85% των συστάσεων του DAC και της εξολόγησης ομοτήμων της εφαρμόζεται είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου. Δηλαδή όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα αυτών, αυτής της για να κάνουν κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές. Λάβατε και την παρουσίαση ενός συναδέλφου από την ομάδα μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης ομοτήμων από το Μάιο στον Οκτώβριο του 2018 έλαβε χώρα αυτή η αξιολόγηση έξι χρόνια δηλαδή μετά την τελευταία αξιολόγηση το 2012 σε αυτή την αξιολόγηση ομοτήμων ως συνήθω υπάρχουν δύο εξεταστές εάν θέλετε ε, η Ιαπωνία και ο Καναδάς στην περίπτωση αυτή με επιτόπιες ε, επισκέψεις στο Μάιο τον Ιούνιο, στο Μαλί και στην Βολιβία. Πρόσφατα συμφωνήσαμε ε, να ολοκληρωθεί αυτή η εξολόγηση ομοτήμων στην Επιτροπή μας με μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αντιπροσωπιών υπό την προεδρία του Φέλιξ Σόρτ. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι αυτή η εξελόγηση ομοτήμων, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έλαβε χώρα σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Όχι μόνο προετοιμάζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναπτυξιακής βοήθειας, υπάρχει και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μέσω λοιπόν αυτής της εκλογής ομοτήμων θέλουμε να επηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο και τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ, στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ε, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης ε, για τις δικές σας εργασίες. Θα ήθελα τώρα να σας πω γενικότερα κάποια αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης η οποία αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας, η DAC, και η διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση σχετική του ΩΣΑ έχει εκφράσει την εκτίμησή της ε, για τον πολύ σημαντικό, πολύτιμο ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων, στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναψυξιακής συνεργασίας, είναι το βασικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης ομοτήμων. Αυτό, αξιολογώντας δηλαδή τις πολιτικές, υπάρχει μια γενικότερη εκτίμηση αυτού του ρόλου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 24 Οκτωβρίου είχαμε τη σχετική συνάντηση. Θέλω να επικεντρωθώ τώρα σε τρεις πυλώνας, πυλώνες. Τομείς δηλαδή όπου είχαμε πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι εκεί όπου υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται αλλά είναι εν εξελίξει αυτή η εφαρμογή Και ο τρίτος πυλώνας είναι κάποιοι τομείς όπου πρέπει να λάβουν χώρα αλλαγές με βάση τις κριτές γραμμές ε, ο ΣΑΝΤΑΚ στην αξιολόγηση ομοτήμων. Σε ό,τι αφορά την, ε, το global leadership, τον ηγετικό ρόλο δηλαδή παγκοσμίω, ε, έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την αξιολόγηση παγκοσμίω Δηλαδή, θεωρούμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μεγαλύτερος δωρητής παγκοσμίω, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη βέβαια, ε, προσωπούν 84 δισεκατομμύρια δολάρια προχρόνο, ο μεγαλύτερος δωρητής του ΝΤΑΚ και αυτό είναι αξιέπαινο. Ταυτόχρονα Το 2016 είχαμε 16 δις εκατομμύρια επιπλέον, δισεκατομμύρια επιπλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο δημιουργώντας ε, ε, συμμαχίες ε, παγκοσμίως παγκοσμίω για να φτάσουμε σε κοινέ θέσεις, στην εφαρμογή σε, όλους τους πυλώνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Παρισίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο επίσης δημιουργώντα συμμαχίε για τη συνολική υποστήριξη σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε στη γραμματεία της Διεθνούς Task Force για το TOXTI και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι, συμπροεδρεύει άλλωστε σε αυτήν την Task Force. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανθρωπιστική βοήθεια, το DAC θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε έναν ηγετικό ρόλο, ακολούθησε μια σφαιρική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την, την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στο παρόν πλαίσιο ε, σειράξεων, ε, ένα εύθραυστο περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει και τα ταμεία επίκουσας βοήθειας για να μπορέσει να απαντήσει σε κρίσει για να αποφευχθούν ε, ε, οι προσεγγίσεις ad hoc το δεύτερο, δεύτερο πυλώνα για να κάνει με την αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή βοήθεια, Αυτό αποτελεί μέρο ε, των βασικών ενισχύων τη ΔΑΚ. Οι βασικέ αρχέ, η σφαιρική ε, σύμπραξη για τα ζητήματα αυτά, το ΔΑΚ ε, ε, επενεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσπάθεια που έχει γίνει για να αυξηθεί από την αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή βοήθεια μέσω τη εκτεταμένη χρήση τη δημοσιονομική υποστήριξη. Όπου αυτό χρειάζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 80% ε, της ε, δημοσιονομικής υποστήριξης από τα μέλη του ΝΤΑΚ. Αυτή η αποτελεσματικότητα της ε, δημοσιονομικής υποστήριξης για την βελτίωση της διακυβέρνησης του κράτους δικαίου όλων αυτών των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο και βεβαίως ε, έχουν συμφέρον όλα τα μέλη να μάθουν από την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική υποστήριξη είναι κάτι το οποίο δεν το μοιραζόμαστε ευρύτερα μεταξύ μελών του ΝΤΑΚ. Επίσης, ε, ο κοινό προγραμματισμός και οι συμπράξεις με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς που λαμβάνουν χώρες 65 ε, χώρες βασίζονται στις προτεραιότητες αναχώρα με οικειοποίηση και συμπερίληψη αυτό βοηθάει στην αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας όπως αυτό, αυτή αναλύθηκε στην αξιολόγηση αντικτύπου ε, στην αξιολόγηση ομορτήμων συγγνώμη. Ε, σε ό,τι αφορά την δημόσια ευαισθητοποίηση ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σημαντικός δημιουργώντας δηλαδή και την αίσθηση της παγκόσμιας ηθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουμε να είναι στην, στην πρώτη γραμμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Θέλουμε να πετύχουμε τα SEGs της Ατζέντα του 2030. Θα πρέπει για να συμβεί αυτό οι πολίτες να είναι στο κέντρο της πολιτικής μας για να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Να περάσω τώρα στο δεύτερο set, στο δεύτερο πακέτο συστάσεων εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ενθαρρυντικά βήματα, αλλά μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτά τα επιτεύγματα. Πρώτα, για τι επιχειρησιακέ κριτικέ γραμμέ, υπάρχει μια, ένα, ένα κοινό στρατηγικό όραμα με τα κράτη-μέλη ε, στην επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Κονσένσου για την ανάπτυξη του 2017. Τώρα ήρθε η στιγμή να αναπτυχθούν περαιτέρω επιχειρησιακέ κριτικέ γραμμέ όπως αυτές εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς δηλαδή τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσουν αυτό το consensus επικεντρωνόμενοι στη μείωση της φτώχειας και τη συμβιώσιμη ανάπτυξη. Βεβαίως η συνένεση αυτή, το consensus αυτό ε, δεν αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το γνωρίζουμε αυτό, επικεντρώνεται και στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις γραμμές ε, γύρω από το consensus αυτό ε, να ληφθούν υπόψη για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ε, Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στι ε, δράσει τη. Υπάρχει όμω περιθώριο βελτίωση ε, να αυξήσουμε τι δυνατότητε, τα κίνητρα, τα μέτρα για να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε αυτά τα μέτρα μεταξύ των διαφόρων ε, εμπλεκομένων φορέων. Είναι σημαντικό αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, συμπεριλαμβάνεται επίσης σε αυτή την ε, αξιολόγηση 27% των χρημάτων που προέρχονται από εκεί. Στο πλαίσιο αυτό εμείς συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αρχίσει να δίνει αναφορές και για το θέμα τη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη αξιολόγηση. Τώρα για το περιβάλλον και την αγκληματική αλλαγή. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει με τη σημαντική πρόοδο ε, έτσι ώστε αυτές οι πολιτικές να γραφούν οριζόντια σε όλους τους τομείς, δημιουργία δυνατοτήτων, έλεγχος της ποιότητας, ε, διευκόλυνση σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Το θέμα είναι κατά πόσο μια ρητή στρατηγική, όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο του 2017, ε, μάλλον στην αναθεώρηση του 2012, ε, αν αυτό ε, μπορεί να οδηγήσει στη μια υποστήριξη της γενικότερης εφαρμογής. ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου το DAC αναπτύσσει κάποια στοιχεία ανάλυσης για τη συνέπεια και την ευθυγράμμιση μεταξύ της, της των Παρισίων και της πολιτικής για την ανάπτυξη, θα προετοιμάσουμε λοιπόν μια έκθεση που θα αξιολογεί την ευθυγράμμιση της πολιτικής συνεργασίας ε, για την ανάπτυξη και ε, τη Συμφωνία των Παρισίων όπως θα γνωρίζετε. Δεν είναι όλα τα στοιχεία 100% συνεπή ή δεν ευθυγραμμίζονται με την Συμφωνία των Παρισίων. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θα είναι πολύ σημαντικός. Ένα άλλο σημαντικό σημείο σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες ε, δραστηριότητες είναι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Ξέρω ότι έχουν γίνει συζητήσει εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, είναι ένα θεμελιώδες, ε, με θεμελιώδης διάσταση για την ατζέντα του 2030. Εάν δεν αυξηθεί ε, η κινητοποίηση ε, πόρων ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιήσουμε χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα και αυτή η κινητοποίηση να πάει προς τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Αυτό είναι κεφαλαιόδες. Σε αυτό το πλαίσιο η έκθεση συστήνει να συνεχιστεί η πρόοδος για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω ενός προγράμματος εξωτερικών επενδύσεων, κινητοποίηση επενδύσεων στην Αφρική αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Ε, ενθαρρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση οι προτεραιότητε των ε, γειτονικών χωρών να είναι ε, σωστά στοχευμένε και να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλων ε, Ευρωπαίων DFIs. Αυτή η συνεργασία, αυτή η προσπάθεια συνεργασία είναι για άλλη μια φορά ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην αξιολόγηση. Για την πολυμερή ενίσχυση, ιδιαίτερα εφόσον αυτή ε, αντιπροσωπεύει το 1 τέταρτο περίπου της νολικής βοήθειας βλέπουμε ότι υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν σειράξεις που παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο θελήσαμε λοιπόν να τονίσουμε εδώ την ανάγκη στα πλαίσια του πολυμερούς χαρακτήρα εφόσον το 1 τέταρτο τη ενίσχυση περνάει από, από, από πολυμερεί οργανώσει, να μπορέσουμε να, εξετάσουμε τον αντίκτυπο. Όλοι συνεισφέρουν σημαντικά σε πολυμερεί οργανισμού και για πολλά χρόνια λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση. Ε, Εμεί ω γραμματεία του ΝΤΑΚ, αλλά και ω μέλη τη Επιτροπή που συμφώνησε για την εξελίξη θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η προσθέμενη αξία αυτή αυτού του τύπου προσέγγισης να τονιστεί περαιτέρω για να γίνει σωστή αξιολόγηση. Τέτοιου είδους συστάσεις έχουμε εισαγάγει σχεδόν σε όλες τις αξιολόγησεις ε, ομοτήμων. Για την συνέπεια της πολιτικής για την ανάπτυξη θέλουμε ενίσχυση του PCD, με σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στι πολιτικέ των κρατών μελών στι αναπτυσσόμενε χώρε, πέρα από την ανάπτυξη, για τη συνεργασία για την ανάπτυξη, χρειάζεται μια παρακολούθηση των εκθέσεων των κρατών μελών για τα PCD και βεβαίω δεν χρειάζεται να το τονίσω περισσότερο αυτό. Να τονίσω δηλαδή το ρόλο των PCD σε αυτή την ε, φιλόδοξη ατζέντα που θα μας απασχολήσει στο προσεχές μέλλον τα αποτελέσματα τώρα της αξιολόγησης. Ε, η αξιολόγηση λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα, τις σχετικές πληροφορίες της αξιολόγησης, διαθρώνοντας ε, μια αφήγηση για την χρήση, τη συνεισφορά, ε, σε ό,τι αφορά τα, τα αποτελέσματα αναχώρα και τον αντίκτυπο που υπήρξε εκεί, πρέπει αυτά να είναι πιο προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, εν περιπτώσει. Τέλος, ε, να αναφερθώ και στα δύο, στους δύο τομείς όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα μιλήσω κυρίως για την ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Το 2015-2016 μόλις 27% της ενίσχυσης πήγε, πήγε προς λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είναι μικρό το ποσοστό. σε σχέση με το μέσο όρο του DAC που είναι 40%. Ε, γνωρίζουμε βεβαίως γιατί συμβαίνει αυτό, γνωρίζουμε την ευρύτερη συγκυρία, όμως είπαμε στο DAC ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και η DAC συμφώνησε να κάνει αυτή τη σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επικεντρωθεί δηλαδή ε, στο θέμα της εκρίζωσης της φτώχειας να αυξηθεί λοιπόν η ενίσχυση προ τι ε, λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Πρέπει επίση να ενισχυθεί ο ρόλο συντονισμού, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να πετύχουν του στόχου του 0,7% καθώς και το 0,15% έως 0,2% για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες σύμφωνα με, και με το consensus. Βεβαίως η Επιτροπή μας θεωρεί ότι επόμενη, το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο δίνει την ευκαιρία, μια σημαντική ευκαιρία να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και να εξετάσουμε πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να προχωρήσουν με συνέπεια ε, επικεντρωνόμενες στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να μην μείνει κανείς μόνος, να μην μείνει κανείς πίσω. Και βεβαίω υπάρχει το θέμα των κατάλληλων δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά τη, ε, απλοποιώντα τι διαδικασίες ε, σε ό,τι αφορά τη επιβάρυνση σε επίπεδο αναφορών και δίνοντας μεγαλύτερη δυνατότητα δημοσιονομική στα κράτη-μέλη επιτόπου. Πρέπει βεβαίως να υπάρχει τακτή αναθεώρηση των πόρων έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει κατάλληλε δεξιότητε κατάλληλες δεξιότητες, κατάλληλες, κατάλληλα προσόντα στις κατάλληλες θέσεις. Τελειώνοντας λοιπόν, να πω ότι βεβαίως και γενικότερα είναι εξαιρετικά θετικό το αποτέλεσμα της εξολόγηση αιμοτήμων, αλλά υπάρχει πάντα και η προσδοκία η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει αυτό το ρόλο τον ηγετικό παγκοσμίω στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Η επιτυχία ε, δεν θα μετρηθεί με βάση τα που συμφωνήθηκαν το 2015, αλλά από αυτά που θα επιτευχθούν το 2030. Ευχαριστώ πολύ. Before μία διευκρίνηση πριν δώσω το λόγο στους αδέλφους. Το σκεφτόμουν ακούγοντά αυτή η εξολόγηση ομοτήμων. Είναι για τις δαπάνες των θεσμικών οργάνων ή της κομισιών, όχι των κρατών μελών της δαπάνες. Α, Γιατί στη σύσταση όλο για τα κράτη-μέλη γίνεται λόγος. Α, μιλάτε για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να το τσεκάρω, να το επιβεβαιώσω. Απλά, καλά το είχα καταλάβει λοιπόν. Ποιοι είναι οι συνάδελφοι που έχουν στήσει το λόγο, η Μαρία Χόιμπουχ και η Χάιντι Χάουταλα. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ωραία. Ευχαριστώ έλεγα λοιπόν για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ήδη είχα κάποιες απορίες, βέβαια και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω ερωτήσεις γιατί το κατάλαβα πολύ καλά. Η Κομισιόν δηλαδή εξετάζεται πώς δαπανά, έχει δαπανίσει τα χρήματα. Δύο τομεί θεωρώ ότι είναι σημαντική. Η κατανομή τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, διότι υπάρχουν πολλέ έτσι ε, ορταστικέ και λογικές εκδηλώσεις για το πόσο καλά τα πηγαίνουμε και έπειτα ε, βλέπουμε ότι μόνο ένα κομμάτι ε, πολύ μικρό δείχνουμε αναπτυξιακής βοήθειας στο κομμάτι της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτή τη σχέση μεταξύ Αφρικής εταιρικής σχέσης πλέον μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια νέα σελίδα ε, και αν δούμε τα χρήματα τα οποία το σύνολο δηλαδή ε, είναι η μεγαλύτερη δικαιούχη. Αν δείτε στην Τουρκία ε, τι ποσά δίνουμε, αυτά δεν πηγαίνουν για την αναπτυξιακή βοήθεια. Βλέπω λοιπόν μία αντίφαση εδώ σε σχέση, επαναλαμβάνω, με την νοτίως της Σαχάρας Αφρική, που πιστεύω ότι πρέπει να την προσέξουμε και θέλω να ρωτήσω και την Κομισιό στο μέλλον τι θα κάνει, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει, ώστε στον τομέα ακριβώς ε, τα χρήματα ε, να τα αξιοποιήσει, γιατί ξέρω ότι ε, δύσκολο είναι να αυξηθεί το ποσό. Σε ό,τι δεν αφορά την συνεκτικότητα της πολιτικής, έχω ένα ερώτημα. Είπατε κι εσείς κάποια πράγματα, είπατε ότι έχει να κάνει με την συνεργασία ε, για τα ε, αναπτυξιακά προγράμματα. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι τι κάνουμε στο μέτωπο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά εμείς εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πολιτική προδιαμορφώνουμε. Και νομίζω ότι κάπως ε, υπολείπεται η πολιτική, η συνεκτικότητα της πολιτικής και για το PCT έχουμε τις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε δύο χρόνια ε, εξέδιδε δημοσιοποιήσει αυτήν την έκθεση. Τώρα δεν την ε, ε, εκδίδει πλέον. Έχουμε όμως τώρα τη νέα γεωργική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργική πολιτικής, ε, που έχει εξωτερικές επιπτώσεις. Και σε ό,τι αφορά τη δική μας γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας και νομίζω θα ήταν πολύ πιο εύκολο να είχαμε αυτή την έκθεση της Κομισιόν ώστε με τη βοήθειά της να μπορέσουμε να πούμε το 2015 ήταν έτσι, το 2016 ήταν έτσι, το 2019 και τα λοιπά θα είναι έτσι. Να μπορούμε να βασιστούμε δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε και να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Όμως, εδώ και τέσσερα χρόνια δεν δημοσιοποιείται πλέον αυτή η έκθεση και η ερώτησή μου είναι ότι θα ήταν καλό να έχουμε τα στοιχεία για τα 28 κράτη-μέλη από κοινού και ποιος θα έχει αυτή την εντολή αν όχι η Κομισιόν. Και το άλλο ερώτημα είναι στο μέλλον πώς σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλο πάντων στο λιγότερο την επόμενη επταετία, τι θα κάνει, πώς θα προωθήσει ε, την συνεκτικότητα της πολιτικής ε, στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης. Ε, γάμα Δέλτα έχει κάποιες ιδέες και πώς μπορούμε από κοινού να έχουμε μια συνεκτική πολιτική την επόμενη επταετία που θα μας οδηγήσει σε βήματα πρόοδου. Thank you. Um, um, Ευχαριστώ η Χάιτι Χάουταλα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι αξιολογίες ομοτήμων της ε, ΩΣΑ είναι κάτι που είναι θετικό και έτσι πρέπει να το εκλάβουμε. Εγώ επιφανειακά, έτσι ακροθυγώς, ε, διάβασα τη περίληψη των συστάσεων. Βλέπω όμως πολλές συστάσεις να πηγαίνουν στη διακατεύση με αυτά που εμείς ζητούμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στιάζει δηλαδή στη μείωση της στόχιας, υπό την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι γεωπολιτικές, μάλλον τόσο πολύ γεωπολιτικοί ε, και άλλοι στόχοι που όλοι ζητούν ε, χρηματοδότηση. Και επίσης μια άλλη σύσταση λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί μέτρηση της, ε, των επιδόσεων του προγράμματος για την ισότητα των δύο φύλων και κατά τρίτον μια ευγενική υπενθύμηση που λέει ότι αν δημιουργούνται νέα καταπιστεύματα η ευθυγράμμιση των ε, στόχων με τους στόχους των χωρών τα υπόψη και θα πρέπει το πεδίο να περιορίζεται σε ένα πλαίσιο κρίσης. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται με όλα αυτά. Και το ότι πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα επίσης ε, και να έχουμε ηγετική ε, εμείς θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από το μέσο όρο του 40% τόσα, με 27% που δίνει στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο όλο αυτό που, όλα αυτά που μα είπατε και προς την Κομισιόν έχω επίσης δύο ερωτήσεις. Υπάρχει αυτή η σύσταση για τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα της πολιτικής και πώς επηρεάζει η πολιτική των κρατομελών και της Ένωσης. Με τι μηχανισμούς θα μπορούσε να κάνει παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσει ε, την συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη με τα κράτη-μέλη. Και μια άλλη σύσταση που λέει μια βασιζόμενη αποδείξει και συνολική πανευρωπαϊκή, πανενοσιακή προσέγγιση, βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕΠΑ και της ε, Κομισιόν και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Η Κομισιόν έχει να μα δώσει μια απάντηση. Νομίζω ότι είναι μια μελέτη που όλοι μας θα τη μελετήσουμε σε βάθος και να αντλήσουμε διδάγματα για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Παραδείγματο ευχαριστώ. Γκέρεν και Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που εκπρόσωπος ε, του ΩΣΑ λέει ότι κάνει καλά τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, υπάρχουν τομείς που τα κάνει πολύ καλά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι τομείς, ας πούμε, όταν εσείς επικρίνετε το γεγονός ότι δεν έχει επιτύχει το στόχο του 0,8%. Δεν ευθύνεται η Κομισιόν ε, γι' αυτό, ευθύνονται τα κράτη-μέλη. Και μπορεί κανείς να το διαβάσει θετικά, ότι δηλαδή η Κομισιόν κάνει καλά τη δουλειά της, αλλά και αρνητικά, ότι υπάρχουν καμιά εικοσαριά χώρες, υπάρχουν καμιά εικοσαριά χώρες που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και διαρκώς ε, στέλνουμε στις ελληνικές καλένδες ε, την ε, ε, αποφασιστικότητα όσον αφορά την τελική απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Δεύτερον, διάβασα έτσι διαγωνίω το έγγραφο και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές, ε, η αρχή της διαφοροποίησης. Αυτές οι αρχές, και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί επανέρχομαι διαρκώς στο ίδιο θέμα, είναι όμως πάντα πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια με τρόπο καθαρό και αποτελεσματικό, ε, θα πρέπει να δούμε, να διαγράψουμε από τον κατάλογο τους ενδιάμεσους. Εάν θέλουμε να εκριζώσουμε την φτώχεια, θα πρέπει πραγματικά να βρούμε κάποια λύση. Και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς να δίνει χρήματα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα μέσω των οποίων μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να παραμείνουμε ε, παρόντες όσον αφορά το, τα πολέμηση του AIDS και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα και με το AIDS και με την φυματίωση και είναι χώρες ενδιάμεσες, δηλαδή ενδιαμέσου εισοδήματος. Επίσης, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έχετε εκτιμήσει την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξέλιξη του κράτους δικαίου στις ε, χώρες δικαιούχους. Και οδηγούμε και στην τέταρτη ερώτηση. Όταν η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσες στην, σε μια χώρα Ποια είναι η χώρα που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε όσον αφορά το θέμα αυτό. Γιατί οι ορισμένες χώρες ε, κατήγγυλαν ε, την συμμετοχή στο ποινικό δικαστήριο, ενώ ε, πρόκειται για ε, ένα από τα θετικά που αναφέρονται στο Κοτονού και τις επιθυμίες που αναφέρονται στο έγγραφο του Κοτονού. Υπάρχουν άλλοι εταίροι οι οποίοι ας πούμε ε, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το σεβασμό των άλλων κλπ. Τι γίνεται. Γιατί νομίζω ότι ένας παγκόσμιος leader, ηγέτης, πρέπει να αναλύει και αυτά τα θέματα. Στην ουσία είναι πολλές ερωτήσεις που θέλω να ε, θέσω και μακάρι να είχαμε ολόκληρη τη μέρα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, κάνει ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Επίσης, είναι καλή όσον αφορά το διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, Πιστεύω ότι προς το συμφέρον μας θα ήταν να έχουμε ένα, μια ομάδα προβληματισμού, ένα είδος think tank που θα δει λίγο πιο πέρα, με προοπτική. Η έκθεση επικρίνει το τι κάνει ε, ο ΣΑ. Δεν θα έπρεπε ε, να υπάρχει έτσι μία διαδικασία προβληματισμού ε, και από τη δική του πλευρά. Ευχαριστώ πολύ, Σάρλε. Η Σάρλο Ατζεντίνη. Ναι, πολλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, οι δύο συνάδελφοι ε, είπαν ακριβώς αυτά που ήθελα να πω, άρα παρετούμε. Στη σελίδα 19 της ε, έκθεσης. Λέτε ότι το EIB είναι εκτός ε, από, τις, ε, από την αγορά αυτή. Αλλά ξέρουμε ότι μέσω τέτοιων εργαλείων ε, θα, δηλαδή μέσω χρηματοπιστωτικών, μέσω δανείων και τα λοιπά ε, θα προχωρήσει ε, η βοήθεια. αλλά εδώ δεν τα λέτε και πάρα πολύ καθαρά. Το είπαμε και χτές ότι καμιά φορά αυτή η πολύ διπλωματική γλώσσα ε, μας αφήνει να καταλάβουμε κάποιο μήνυμα, αλλά ε, δεν ε, καταλαβαίνουμε και ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Επίσης, ποια είναι η αξιολόγηση ε, που κάνετε όσον αφορά τα συστήματα δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αν χρειαστεί να δώσουμε περισσότερα χρήματα και για τον ιδιωτικό τομέα τότε θα πρέπει να ξέρουμε να έχουμε περισσότερες γνώσεις ε, ναι, είναι γεγονό ότι πανάκια δεν υπάρχει. Τέτοιου είδου λύσει δεν υπάρχουν. Ούτε ο ιδιωτικό τομέα λοιπόν είναι πανάκια. Ε, και καμιά φορά περιμένει κανείς ότι χρηματοδοτώντας τον ιδιωτικό τομέα ε, θα ε, διονγκωθεί το κέρδος ή θα υπάρχει προσεκτικότητα ή επιστροφή, αλλά καμιά φορά δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικά, γιατί μιλάμε για δημόσια χρήματα. Πιστεύετε ότι η Κομισιόν στην αναπτυξιακή πολιτική μετράει καλά ε, την μετακίνηση των, ε, των πόρων ε, και την προσθετικότητα κλπ. Επίσης, κάποια εξειδικευμένα εργαλεία ή εργαλεία ειδικού στόχου και σκοπού. μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα επιπλέον. Και τέλος, στρεφόμενοι προς την Κομισιόν. με ποιο τρόπο θα αντικατοπτριστούν αυτά τα νέα διδάγματα στα νέα προγράμματα. θα μας ε, ε, μιλήσει και προς του Κόγκορντ και μετά της ε, Κομισιόν. Ίσως κάποιος να πει και στον κύριο Επίτροπο ότι δεν θα ξεκινήσουμε ίσως ακριβώς τις 4, 5-10 λεπτά και αργοπορία θα έχουμε. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, αλλά σίγουρα Κάποιες οι οποίες απευθύνονται από την Κομισιόν θα απαντηθούν από αυτήν. Εγώ θα προσπαθήσω να καλύψω αυτά τα οποία ίσως είναι πιο ενδιαφέροντα για την Επιτροπή σας. Ναι, πρώτα απ' όλα για το PCD είναι σημαντικό νομίζω να υπογραμμίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε τη σημασία του PCD δεν έχει να κάνει μόνο με τις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας, αναπτυξιακής συνεργασίας θέλουμε να πάμε πέρα από το να μην κάνουμε κακό στις άλλες πολιτικές. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο σφαιρική προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές, σε όλους τους θεματικούς, ε, στις θεματικές ενότητες. Έτσι λοιπόν όντω το PCD εγγράφεται στα πλαίσια μιας σφαιρικής προσέγγισης, συνολικής προσέγγισης για την ανάπτυξη. Χρειάζεται παραδείγματος χάρη ευθυγράμμιση μεταξύ των 3 D. Διπλωματία, άμυνα, ανάπτυξη. Και αυτός ο κατακρεματισμός που υπάρχει, αυτή η ασυνέπεια αν θέλετε, σχετίζεται και με το πώς αναπτύσσουμε τις δημόσιες πολιτικές μας, ε, στις πρωτεύουσές μας. Θέλω να είμαι σαφής λοιπόν. Βεβαίως και θεωρούμε ότι το PCD είναι μια υποχρέωση για όλες τις πολιτικές πέρα από την ε, αναπτυξιακή, αναπτυξιακή συνεργασία. Τώρα είπε ο κύριος Ότολα μια σειρά από πράγματα, τα πιο πολλά νομίζω απευθύνονται στην Κομισιόν, αλλά κάτι που θα ήθελα να πω είναι το εξή. Οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και ε, το πώ επικεντρωνόμαστε στην εκρίζωση τη φτώχεια. Αν ακολουθήσουμε απλά τι τάσει που υπάρχουν, εγώ είμαι στη γραμματεία της DAC ε, και πέρα από το ODA. Αν ακολουθήσουμε τις τάσεις βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι θετικές ε, για την εφαρμογή των SDGs διότι το θέμα δεν είναι μόνο η κατανομή των πόρων προς λιγότερο αναπημένες χώρες που πρέπει να αυξηθεί αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα πολύ περίπλοκοι μηχανισμοί όπως το lended finance αυτό συνδέεται και με το ρήμα της Προέδρου. Όλες οι ξένες άμεσες επενδύσεις, όλα αυτά πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση τελικά. Μεγάλες δυνατότητε, σωστοί μηχανισμοί, κινητοποίηση, η οποία είναι λυπή στα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω δημόσιων πρωτοβουλειών, σε ό,τι φορά όμως το 7% είναι μόλις 27% μάλλον το τι πάει στις ε, ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Πρέπει να κάνουμε να βελτιωθούμε πολύ. Είμαστε εδώ πιο πίσω και από το ODA. Στον ιδιωτικό τομέα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι, οι, οι άμεσε ξένε επενδύσει. Ένα πολύ μικρό <laughs> ποσοστό πάει προ τι έθραυστε χώρε. Όπου 80% των πιο, πλού, των πιο φτωχών θα ζουν εκεί μέσα στο 2030. Ε, πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για να εκριζώσουμε τη φτώχεια και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση των έστραφτων χωρών. Αν όμως αφήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει μια τάση χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση, δεν θα τα καταφέρουμε. Χαίρομαι λοιπόν που διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη παίρνουν πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό, προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες τους με ε, τις αρχές του ΟΣΑ και του ΝΤΑΚ. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να καλυφθούν κάποιες ασυνέπειες που υπάρχουν. Αυτή η ιδέα του ότι θεωρούμε ακόμα επιλέξιμη βοήθεια για, το, για τα ορυκτά καύσιμα στις χώρε, χώρες, αναπτυσσόμενε χώρες, το θέμα των εμβασμάτων. 3-3 ε, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Όμως το κόστος συναλλαγής είναι συχνά έως και 20%. 1% πιο κάτω να πηγαίναμε σε ό,τι αφορά τα εμβάσματα, στο πώ φορούμε τα εμβάσματα, θα, θα μείωνε κατά 30 δις το ποσό. Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν δεν είναι απλά κάτι το οποίο το λέμε ως ρητορική. Πρέπει ε, να παίξουμε το ρόλο μας ως ε, ε, ρυθμιστική αρχή, ως νομοθέτης, ως νομοθέτες. Χαίρομαι που αυτό το έχει ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανησυχίες της και ελπίζω πλέον ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, στα πλαίσια και το πολιτισμό του δημοσιονομικού πλαισίου ε, θα αναπτύξουν περαιτέρω αυτήν την ατζέντα. Κάτι ακόμα δεν μπορώ βεβαίως να απαντήσω σε όλα. Να προσθέσω όμως κάτι σε σχέση με τα ερωτήματα για την μετάβαση και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Είναι αλήθεια ότι οι χώρε μέσω εισοδήματο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια και τι ανισότητε. Και οι δωρητέ, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο θεσμό και τα κράτη-μέλη, πρέπει να γνωρίζουν ότι βεβαίω πρέπει να επικεντρωθούμε και να δώσουμε προτεραιότητα στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε ε, μια χώρα η οποία περνάει από το καθεστώ τη λιγότερο αναπτυγμένη χώρα σε ένα άλλο καθεστώ. Πρέπει όμω βεβαίω να βασιζόμαστε σε αποδεικτικά στοιχεία, σε δεδομένα. Διότι υπάρχει μεγάλη υποκειμενικότητα και ένα ιδεολογικό χαρακτήρα ό,τι αφορά το πέρασμα από τη μια κατηγορία στην άλλη, ιδιαίτερα από τι χώρε τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζω ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε την επαφή με τι χώρε τη Λατινική Αμερική. Εξακολουθούν να πρέπει να κάνουν πολλά για να αντιμετωπίσουν τι ανισότητε και τη φτώχεια. Ταυτόχρονα αυτό που ζητάνε ε, είναι περισσότερο συνεργασία. Αυτή λοιπόν η έννοια της μετάβασης αντί για το άμεσο πέρασμα σε μια άλλη κατηγορία είναι, το, είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια μετάβαση δηλαδή. Ακόμα όμως και το πέρασμα σε μια άλλη κατηγορία, προβιβασμό αν θέλετε, έχουμε κάνει μια δουλειά, μπορούμε να τη μοιραστούμε και μαζί σας, έχει γίνει μελέτη για το τι συμβαίνει όταν μια χώρα προβιβάζεται και δεν είναι πλέον λιγότερο αναπτυγμένη χώρα. Αυτό που συμβαίνει άμεσα είναι ότι υπάρχει αμέσω έλλειψη ε, πόρων για την εκπαίδευση, για την υγεία και αυξάνεται το χρέο. Πρέπει λοιπόν μεταξύ των δωρητών και των αναπτυσσόμενων χωρών να υπάρξει μια σύμπραξη για να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο σε ό,τι αφορά του οικονομικού πόρου, γνωρίζοντα ότι καθώ μια χώρα αλλάζει επίπεδο, ε, πολλά πράγματα μπορούν να ε, τακτοποιηθούν με διαφορετικούς, από διαφορετικούς, ε, διαφορετικούς οικονομικούς πόρους, ε, χρηματοδότηση για το κλίμα, χρηματοδότηση για κοινωνικούς λόγους, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Θα σας δώσουμε μάλιστα και στοιχεία για το τι συμβαίνει ε, στις χώρες αυτές. Τώρα για την Κίνα και τον ΤΑΚ. Θα μπορούσα να σας μιλάω όλο το απόγευμα για το θέμα αυτό, όπως φαντάζεστε. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι δεν αφορά μόνο τα χρήματα αυτό. Αφορά τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα. Και πραγματικά χαίρομαι που εργάζομαι με χώρες που σκέφτονται όπως εμείς, όπου όλο το έργο για την αναπτυξιακή ενίσχυση βασίζεται σε αρχές ε, και στην αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιο να είναι μέλο του DAC για να έχει μια σωστή προσέγγιση για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και βεβαίω συνεργαζόμαστε με την Κίνα και με άλλε αναδυόμενε οικονομίε για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία, μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και να επικεντρωθούμε όλοι ε, στα πιο σημαντικά. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, για αυτό που είπατε για το ρόλο του EIV. Εδώ Προφανώς και ο Φέληξο το γνωρίζει. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε απαιτεί συνένεση. Το DAC δηλαδή εργάζεται σε ένα συνενετικό ε, πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η γλώσσα, η διατύπωση είναι πάντα προϊόν διαπραγμάτευσης. Όμως αυτές τις παραγράφους ε, δεν υπάρχει λάθος. Έτσι. Μην, μην, κάνετε λάθος. Εδώ ζητούμε να αναλυφθεί δράση για μεγαλύτερο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με προσανατολισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των, των τομέων προτεραιότητας. Υπάρχει ένα προγραμματισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητες και πρέπει από εκεί και πέρα και το, το, το ε, των επενδύσεων να είναι συνεπές με αυτόν τον προγραμματισμό. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αν το EFSD επεκταθεί ως προς το δημοσιονομικό με πολλά δις, γιατί αρχικά ήταν για τα πιο ευάλωτα κράτη, εκεί που δεν μπορούσαν να φτάσουν τα χρήματα. Γι' αυτό το συστήσαμε και το, συγκροτη... το ονομάσαμε EFSD-SYN είναι εδώ και ο συνεισηγητή, ο κ. Γκέρενς. Και φαντάζομαι ότι αυτό τα λάβουμε υπόψη μας να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Τώρα πέρασε τώρα στο Κόνκορτ, τη ΜΚΙΟ, ε, που υπομονετικά περιμένουν. Ο Τζόναθαν Μπίγκερ είναι το όνομά σας. Συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Αν μπορείτε όμως σύντομα να μας πείτε δύο πράγματα. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση που δίνεται λόγο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ε, των ΜΚΟ για ε, ανθρωπιστική βοήθεια 28 ενώσεις 24 διεθνή δίκτυα. 2.600 ΜΚΟ συνολικά εκπροσώπου, της Jonathan Bigger λέγομαι. Είμαι μέλος της Concord. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον ΩΣΑ για την επικοδομητική και κριτική αυτή ε, αξιολόγηση. Την καλωσορίζουμε, συμφωνούμε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί που μας κάνουν περήφανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την τελευταία έκθεση και μετά όπως αυτή η συνένεση, την ανάπτυξη, το κοινόρμα που είπατε κι εσείς, υποστήριξε επίσης των χωρών εταίρων τη βιώσιμη ανάπτυξη και προώθηση ε, της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Συμφωνώ λοιπόν ε, με πολλά και εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε κάποιες επιλεκτικά από τις συστάσεις που ανταποκρίνονται και στη βασική έκκληση των δικτύων των ΜΚΟ. Τα σχόλιά μου τα κάνω επειδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε την αποφασιστική διαφορά στο ό,τι αφορά του ΩΣΑ για το σχεδιασμό του εξωτερικού εργαλείου του προσεχούς πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Νομίζω ότι ε, θα συζητήσετε τροπολογίες αργότερα σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει σοβαρά υπόψη σε αυτές τις συστάσεις. Έχουμε κάποια παραδείγματα όπως την κλιματική αλλαγή. Επανέρχονται λοιπόν κάποιες συστάσεις. Έλειπαν από μια συνολική αντιμετώπιση στο πλαίσιο του πολιετούς Άρα τώρα έχουμε την ευκαιρία, η στόχη βασιμής ε, ανάπτυξη την επόμενη φορά, στο προσεχές πι να είναι πιο πλήρης αυτή η στόχη. Τέσσερες σύντομα στάσεις θα σχολιάσω για το τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει τώρα. Και απευθύνομαι και στους βουλευτές που διαπραγματεύονται τώρα. ώστε οι συστάσεις που ακούσαμε να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Πρώτο, για επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των συστάσεων. Αυτή είναι μια πρόταση του ΩΣΑ. Αυτό το εξωτερικό εργαλείο θέλουμε να εστιάζει στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και εκρίσωσης της φτώχειας. Πρέπει να προσθεθούν στην ατυχή έλλειψη ε, αυτών των δηλαδή να συμπληρωθεί ε, το αρχικό κείμενο που ε, τυχώς δεν περιελάμβανε. Σε αυτό συμφωνούν και οι χώρες μέλη και το Κοινοβούλιο. Και επίσης η έλλειψη της ε, συνεκτικότητας πολιτικής δεν θα καλυφθούν μόνο με αυτό το εργαλείο, αλλά και με μια ολόκληρη διαδικασία θα θέλαμε να ακούσουμε τις προτάσεις Κομισιόν Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, για μελισσότερη συνεκτικότητα. Αλλά λίγα θα γίνουν αν το SDSR παραμείνει να μην είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. Μας είπε και ο Σάκη, αυτό είναι το δεύτερο, 43% στις χώρες μεσαίου Στο εισοδήματο και το 27% στι πιο φτωχές ή πιο ευάλωτε. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Για μας είναι μεγαλύτερη και τελευταία ευκαιρία πριν από την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι τώρα Επίσης, ε, σε ό,τι την πρώτη συνένεση για την ανάπτυξη, 0,1 ή έως 0,2 έπρεπε να πάει λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από το 2015 δεν έχει εκπληρωθεί ο στόχος αυτός και νέα ημερομηνία το 2030. Πολύ περιθωριακά έχουν βελτιωθεί οι συνεισφορές προς αυτές τις χώρες. Είμαστε στο 0,11%. Πώς θα γίνει πράξη αυτή η δέσμευση. Αυτή τη στιγμή δύο πράγματα πρέπει να γίνουν και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνεί μαζί μας. Η κατηγορία 6 στο νέο ΠΔΠ πρέπει να είναι 92% και πρέπει να υπάρχουν βασικές δεσμεύσεις για το 0,2% προς λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε στα άρθρα του εργαλείου. Και συμμετοχική διαδικασία για όλους. Ένα νέο σχέδιο δράση για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες. Τρίτον, στάσει του όσα μας προειδοποιούν και μας λένε ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα άτομα, στους ανθρώπους. Το βασικό είναι αυτή η επενδύση την ανάπτυξη, είναι γύρω στο 11%. <clears throat> για 20% είναι ο φιλόδοξος στόχος που νομίζω ότι πρέπει να λέγεται και στο ίδιο το σώμα του κειμένου και όχι μόνο στο προήμιο. Οι ανθρώπινε εξέλιξει, η ανθρώπινη μάλλον εξέλιξη βασίζεται στην ανάπτυξη τη υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και ε, άλλο το φύλλο. Είναι διαφορετικά θέματα αυτά. Χρειάζονται και χωριστοί στόχοι που πρέπει να εντοπιστούν σωστά. Και τα σημεία αναφορά στα benchmarks δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε γιατί μα ε, βοηθούν. Και το τελευταίο σημείο στην Επιτροπή σας θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σοβαρά τα περί μεικτή χρηματοδότησης ε, blended finance. Το 8% για την ΕΤΕΠ συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε και στοιχεία για τι γίνεται με αυτό το μείγμα, αυτό το, το blending. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε περισσότερα στοιχεία και μετά να δαπανηθούν περισσότεροι πόροι και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις βασικές προτάσεις που συζητάτε. Αυτό προτείνεται, είναι πολύ καλό και μακάρι να γίνει. Όμως, σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα που είπατε, δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού. Ελπίζω απόψε να φροντίσετε να ξαναμπούν σε αυτόν τον κατάλογο εξαίρεση ή αποκλεισμού. Και για το πι στην ε, αξιολόγηση λέγεται ότι υπάρχει μια γενναιόδορη μεν ανταλλαγή με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχετική στρατηγική. Δηλαδή να δίνουμε κατά αποκοπήν ποσά σε ένα φορέα μόνο για ένα συγκεκριμένο θέμα είναι μια καλή στρατηγική. Όπως βλέπουμε για το φύλλο, διπλασιάζει το διοικητικό κόστος. Αυτό το λέει αξιολόγηση ομοτήμου. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Και αυτή η spotlight ίσχυτη, αυτή η πρωτοβουλία φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε ε, στο επόμενο θέμα μας, στις τροπολογίες. Στην επόμενη συνέντευξη θα το δούμε. Έχουμε τον Φέλιξ Φερνάντεθ Σό. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον ε, Ζωσ ε, και τους υπολείπους. Είναι η τρίτη ε, αξιολόγηση αιωμοτήμων. επισκόπηση. Έχω κάνει άλλες ε, δύο και εδώ έχουμε την τρίτη όσον αφορά την μετακίνηση πόρων και χρημάτων. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλή συνεργασία με τον Καναδά και την ε, Ιαπωνία ε, και εμείς έχουμε ε, συνηθίσει πια να κάνουμε μια σειρά από ερωτήσεις, μερικές πιο απλές, μερικέ πιο περίπλοκες, πώς κάνετε, πώς λειτουργείτε, με ποιο τρόπο ακριβώ. Νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν, ε, γιατί ε, κατανοούμε και εμείς οι ίδιοι καλύτερα τι κάνουμε, μοιραζόμαστε με τους άλλους τις αρχές μας και τις αξίες μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ σημαντικά και για την τωρινή και την μελλοντική μας ε, δουλειά. Κοινό προγραμματισμό ας πούμε, ε, υποστήριξη, δημοσιονομική υποστήριξη και συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών ε, πολιτικών. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στα σχόλια που έκαναν και οι βουλευτές και ο από το Κόγκορντ και ο Ζόρζ. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει ε, να ξεκαθαρίσουμε τα LDCs και την Αφρική γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για λιγότερο αναπτυγμένε χώρε που μπορεί να είναι στη Λατινική Αμερική, μπορεί να είναι στην Ασία, δεν είναι μόνο η Αφρική. Δεύτερον, ε, εάν ε, έχει κανείς ε, ας πούμε μια μεγάλη κρίση ε, στη γειτονιά σας σε χώρες μεσαίου εισοδήματος αυτό σημαίνει ότι κάνουμε επενδύσεις όχι προς τις χώρες αλλά στις χώρες προσπαθούμε να βοηθήσουμε ας πούμε την Τουρκία να ε, αντιμετωπίσει την, ε, τους ε, μετανάστες πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφος της. Επίσης έχουμε γειτονιά σε περιφέρεια με χώρες υποδιεύρυνση και επομένως και εσείς θα πρέπει να σκεφτείτε τώρα εάν θέλετε ε, πραγματικά να φύγετε από τις ε, χώρες ε, μικρού μεσαίου εισοδήματος. Ο, ο κύριος είπε ότι ήδη έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τη διαφοροποίηση και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο στις χώρες μεσαίου εισοδήματος στη γειτονιά μας και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δουλέψει τόσο πολύ με τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γιατί δουλέψαμε πολύ με την Ουκρανία, με την Τουρκία, με την Τινησία κλπ. Δεύτερον, η εστίαση στη μείωση της φτώχειας και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ε, εκ πρώτη όψεω ε, η επικέντρωση στην ε, εκρίζωση της φτώχεια θα σήμαινε ας πούμε επικέντρωση στον, στους φτωχούς αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι και όπως είπε και ο, ο Ζόρζ αν δουλέψουμε εφιώς με χώρες μεσαίου εισοδήματος τότε θα βελτιωθεί η κατάσταση ναι, γιατί σε αυτές τις χώρες μπορεί να έχουμε τη ε, τον μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά κλιματική αλλαγή, όσον αφορά μετρίαση κρίσης κλπ και ε, ε, με ποσοτικούς ε, όρους είναι πιο εύκολο να δουλέψει κανείς με χώρες ενδιάμεσου εισοδήματο παρά με φτωχές χώρες αλλά και αυτό περιλαμβάνεται και στο θεματολόγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα από όλες τις πλευρές. Τρίτον, είχαμε μια μακρά συζήτηση και στον ΩΣΑ, στην ΤΑΚ, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Ε, έγιναν συζητήσεις, θα γίνουν κι άλλες. Και εμείς σαν Κομισιόν προσπαθήσαμε ε, να ε, πούμε, αλλά αυτά είναι τα μηνύματα και από τον ΩΣΑ, ότι ε, πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο και τις προτεραιότητες των χωρών και τις ανάγκες τους και όχι να επιβάλλουμε εμείς αυτό είναι ο σωστό ε, προγραμματισμός και αυτή είναι η συνεργατική αντιμετώπιση. Και εμείς προτείναμε και μία ανοιχτή αρχιτεκτονική για το μελλοντικό ESD και στο δεύτερο βήμα του EFSD να δουλέψουμε ακριβώς με τις ε, ε, επενδύσεις ε, και προς τα πού θα πρέπει να πάνε, γιατί δεν πηγαίνουν μόνος τους αυτές οι επενδύσεις, πρέπει να τις προγραμματίσουμε, να δούμε ε, πώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Μαλί, πώς μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες επενδύσεις στην Μιανμάρ. και ο Ζόρζο και ο συνάδελφος από την Concord ε, ε, είπαν πώς μπορούμε να απομακρυνθούμε, ε, με ποιους τρόπους θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίω θα πρέπει να σκεφτούμε το EIS. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη περίοδο. Δουλεύουμε σκληρά για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε στην ε, συνολική εικόνα και το θεματολόγιο του 2030. Και όχι μόνο, αλλά και το, ε, τις αποφάσεις ε, του Παρισιού για το κλίμα κλπ. και να το κάνουμε δημιουργώντας, χρησιμοποιώντας τις πραγματικές μας ικανότητες ε, και την διάθεση συνεργασίας με τις άλλες χώρες και τους εταίρους μας. Και αυτό βεβαίως ε, προϋποθέτει μια ε, πολυμερή προσέγγιση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζώσο και την Κάρη για την συνεργασία τους, γιατί πολλά μας δίδαξαν, μας έμαθαν καινούργια πράγματα και τώρα βεβαίως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας και να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φέληξ για τις εξηγήσει που μας έδωσες. Δεν χρειάζεται να ε, ε, ξανάρθετε. Νομίζω ότι πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Ε, η αξιολόγηση από αμοτήμους ε, ήταν ενδιαφέρον να το να την ακούσουμε και τα επόμενα χρόνια θα παρακολουθούμε. Και για τα νέα μέλη της Επιτροπής νομίζω ότι καλό θα ήταν να, ξέρουν ποια είναι τα πολιτικά ζητήματα. um, so thank, thank Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και που ξαναήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα παλιά σας λιμέρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Concord, ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Στυλιανίδης ε, και λυπούμε πολύ που σας ε, ανάγκασα να περιμένετε για 15 λεπτά. Okay, colleagues, we've Λοιπόν, συνάδελφοι, αργήσαμε και να ξεκινήσουμε. Όσοι φεύγουν από την αίθουσα, σας φύγουν ε, ήσυχα. Περνάμε σε ένα σημαντικό ζήτημα, το σημείο 22 της Μέσης Διάταξης, το πρόγραμμα εργασιών και επιχειρησιακή στρατηγική της Ευγενικής Διευθυνσής ΕΚΟ για το 2019. Χαιρόμαστε που είναι εδώ ο Επίτροπος για άλλη μια φορά μαζί μας, ο Χρήστος, ο Χρήστος Τηλιανίδης. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα έρθει να μας παρουσιάσει το επικοινωνιακό πρόγραμμα, κύριε Επίτροπε. Μου φαίνεται σαν χθε που αρχίσαμε τη συνεργασία μας. Τώρα βεβαίως είτε έχουμε Brexit είτε όχι, όπως και να έχει, είναι η τελευταία φορά που εξετάζουμε το ετήσιο πρόγραμμα. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα σα δούμε βεβαίω. Ε, πριν ε, τελειώσει η θητεία του Κοινοβουλίου, θα σα πούμε και στην Ολομέλεια και ξανά στην Επιτροπή μα, θα έχουμε ευκαιρίε. Συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τη Ρουμανική Προεδρία για τι προκλήσει που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση. Μιλήσαμε για την κρίση αυτή ε, που διαιωνίζεται αλλά και τις πιο καινούριε κρίσεις ε, στη Βενεζουέλα, στην Ιεμένη πολλά ε, θα είχα να πω, αλλά προτιμώ να σα δώσω το λόγο και να δώσουμε ερωτήματα μετά. Είστε πάντα σαφεί εσεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Λίντα, αξιότιμοι συνάδελφοι, φίλοι. Καλή χρονιά. Παρότι είναι προχωρημένος ο Γενάρης. Είναι πάντα πάντως ευχάριστο να επανέρχομαι εδώ, να έρχομαι ξανά εδώ στην οικογένειά μου. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας. Είναι σημαντικό λοιπόν που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Γνωρίζετε ότι οι συμβουλές σας, η υποστήριξή σας ήταν ε, ανεκτήμητης αξίας για μένα τα τελευταία χρόνια. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την δέσμευσή σας αλλά και για τον ηγετικό σας ρόλο. Αγαπητοί φίλοι, η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, εγώ ως Επίτροπος έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα όλοι μαζί, ανά τον κόσμο, στη Συρία, στην Ιεμένη, στο Μιαμάρ, στη Μιαμάρ μάλλον, στην περιοχή του Σαχέλ, στη Βενεζουέλα. Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα. Εσείς υποστηρίξατε το πιο σημαντικό μέρος του έργου μας. Να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα ε, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση σε δύσκολες καταστάσεις. Το να βάλουμε τέλος στην βία που βασίζεται στο φύλλο, σεξουαλική κακομεταχείριση, ε, σε επίκους καταστάσεις, δημιουργία ανθεκτικότητας και προστασίας ε, για τους μετατοπισμένους ανθρώπους, δημιουργία πιο ισχυρών ε, συμπράξεων μεταξύ ε, των εργασιών μας στον ανθρωπιστικό, στον ανθρωπιστικό και στον πολιτικό τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Πετύχαμε πολλά, αλλά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Αλλά η πολιτική μου φιλοσοφία είναι η εξή. Καθώς αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, ταυτόχρονα δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε και για τις επιτυχίες μας. Θα ήθελα να αφερθώ σε τέσσερις από αυτές τις επιτυχίες. Επιτυχίες ε, που θα συνεχίσουν να αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες και γι' αυτό το έτος. Πρώτον, η εκπαίδευση σε κατάστασεις επίγουσας ανάγκης. Χάρη στην υποστήριξή σας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, καταφέραμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πρώτη δύναμη σε αυτή τη δράση. Τη εκπαίδευση δηλαδή σε απίκου καταστάσει. Μέσα σε τρία χρόνια έγινε αυτό. Φέτο μάλιστα ε, το 10% του ανθρωπιστικού μας ε, προπολογισμού θα πάει σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης ε, σε επίκουσε καταστάσεις. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό κατά τη διάρκεια τη θητεία μου. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για την πολιτική αλλά και τη δημοσιονομική σα υποστήριξη. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως αυτήν την Επιτροπή. Διότι με υποστηρίξατε από την αρχή για τη δημιουργία αυτού του πρώτου ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για το θέμα της εκπαίδευσης, της παιδείας ε, σε επίγους καταστάσεις. Το ζητήσατε εσείς πριν από 18 μήνες και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και πέρυσι το πετύχαμε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν αποτελεί μόνο μια επένδυση ανθρωπιστική. Είναι μια επένδυση στην ειρήνη. Είναι μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον. Δεύτερη προτεραιότητα. Η βία για λόγους φίλου. Η δεύτερη επιτυχία μας έχει να κάνει με αυτήν την, αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου σε επίγουσε καταστάσεις, όπου η εκπαίδευση βεβαίως παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πρόσφατα αφήσαμε την πρώτη θέση στον Καναδά στα πλαίσια του call to action για την προστασία ε, από τη βία που βασίζεται σε φύλλο. Ο Καναδάς όμως ε, εδώ έρχεται να κληρονομήσει μια πρωτοβουλία με 18 νέα μέλη, ε, εξαιρετικά έτσι, ανθούσα πρωτοβουλία, 82 μέλη συνολικά κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Συμμετέχει πλέον και η Νιγηρία, η Δημοκρατία του Κονγκό. Το θέσαμε και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το θέμα. Βεβαίω το γεγονό ότι παραδίδουμε τι κοιτάλε στον Καναδά δεν σημαίνει ότι εμεί πλέον δεν ασχολούμαστε με αυτό. Εμεί θα εξακολουθούμε να πρωταθλητέ ε, στην ε, μάχη κατά τη βία ε, που βασίζεται στο φύλλο. Τρίτον, το θέμα του έμπολα. Μπορούσαμε το 2018 να αντιμετωπίσουμε δύο συνεχόμενα, συνεχόμενες επιδημίες ε, του ιού έμπολα στον Κονγκό. Κινηθήκαμε γρήγορα, συντονισμένα και ουσιαστικά εφαρμόσαμε τα διδάγματα του 2014. Ήταν πολύ ε, επώδυνη αυτή η εμπειρία πριν από κάποια χρόνια στη Δυτική Αφρική. Τώρα όμως, χάρη στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, κινηθήκαμε διαφορετικά Παραδείγματο χάρη κινητοποιήσαμε τα ευρωπαϊκά σώματα, ιατρικά σώματα. Ξέρετε ότι αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεγάλες ε, υγειονομικές ε, επίγουσες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει, ε, αποδεικνύει μάλλον, ότι ποτέ πλέον δεν υποτιμούμε τον ιό έμπολα. Και ευχαριστώ που από κοινού δημιουργήσαμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα η δεύτερη επιδημία έμπολα επηρεάζει τις πιο ε, ανασφαλείς ε, περιοχές, ε, τις πιο ασταθείς περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας, αυτή η επιδημία θα πάρει μήνες για να μπορέσει να ελεγχθεί. Οπότε καταπολεμούμε όχι μόνο αυτήν την ε, ασθένεια, καταπολεμούμε και τους περιορισμούς ασφαλείας και πολεμάμε απέναντι στον χρόνο ουσιαστικά, τρέχουμε με αντίπαλο το χρόνο, έχουμε καταφέρει ήδη να μην αφήσουμε τον ιό να περάσει τα σύνορα στις γειτονικέ πόλεις. Είναι ήδη αυτό επιτυχία, αλλά δεν πρέπει η πρόοδος να συγχαίεται με την εκρίζωση. Ο έμπολα παραμένει προτεραιότητά μας, πρέπει να επαγρυπνούμε και δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ε, εφησυχάσουμε. Τέταρτον, η αποτελεσματικότητα στις εργασίες μας, στον ανθρωπιστικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, το πώς παραδίδεται αυτή η ανθρωπιστική ενίσχυση είναι ορισμένε φορές το ίδιο σημαντικό με την ίδια την ενίσχυση, με την ίδια τη βοήθεια. Και έρχομαι εδώ στο θέμα της ε, ε βοήθειας της ε, συνδρομής σε ρευστό. Το ρευστό δίνει ευελιξία, δίνει επιλογές και έχει να κάνει και με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που βοηθάμε το ρευστό αυξάνει και την αποτελεσματικότητα. Μειώνει το γενικό κόστος. Αυτό είναι σημαντικό. Το είδαμε αυτό ιδιαίτερα στην Τουρκία και στο Λίβανο. Επίσης ταυτόχρονα αυξάνεται η καθαρή αξία της συνδρομής μας, της βοήθειάς μας, μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερα καλά πράγματα με λιγότερα χρήματα διαθέσαμε 35% της ενίσχυσής μας της ανθρωπιστικής το 2018 μέσω μετρητών. Και αυτό θα συνεχιστεί και το 2019. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανθρωπιστική βοήθεια σε ρευστό έχει μια άμεση και βιώσιμη επίπτωση, αντίκτυπο. Είδαμε τα θετικά αποτελέσματα παντού, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Αφγανιστάν, στην Ελλάδα, ε, στη Σομαλία και αλλού γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ανάγκε ανθρωπιστική βοήθεια παγκοσμίω αυξάνονται κάθε χρόνο. Δυστυχώ η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα, αρκέσει, δεν θα αρκεί ποτέ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Για να πετύχουμε μια σταθερή, ε, ένα σταθερό, ε, βιώσιμο μέλλον με ευημερία, θα πρέπει όλοι να χτίσουμε πάνω σε μια βάση ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εργαστεί για να ενισχύσουμε την σχέση μεταξύ ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού τομέα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις βάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτή θα είναι και η προτεραιότητά μας και φέτος. Βεβαίως, όπως πάντα, αναμένουμε την υποστήριξή σας σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Θα ήθελα τώρα με την ευκαιρία που μου δίνεται ε, να συζητήσουμε τις περιφερειακές προτεραιότητες μας. Δυστυχώς ε, το 2019 κληρονόμησε πολλές από τις ανθρωπιστικές τραγωδίες, ε, τραγωδίες του περασμένου έτους Συρία, Ιεμένη, Νότιο Σουδάν, περιοχή του Σαχέλ, τη λίμνες του Τσάντ, Μιαμάρ, Βενεζουέλα, Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα. Να ξεκινήσω από τη Συρία. Η σύραξη έχει κάπως περιοριστεί σε κάποιες περιοχές. Όμως, οι τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν. Σε αυτήν την διαλυμένη χώρα, οι δράσεις μας σώζουν ζωές και προσπαθούμε επίσης να επαναφέρουμε την ελπίδα, την προοπτική. Γνωρίζω ότι το Μάρτιο θα λάβει χώρα η τρίτη διάσκεψη των Βρυξελών για τη Συρία με την Φεντερίκα και άλλους επιτρόπους. Ξέρετε ότι εξακολουθούμε να είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής και στην κρίση της Συρίας, σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν Σύριοι πρόσφυγες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε το έργο του νέου ειδικού επεσταλμένου των ΗΕ, του Γκέρ Πέντερσεν, και, και βεβαίως είμαστε δεσμευμένοι προς το διάλογο. Θέλουμε μία κοινώ αποδεκτή λύση για να μπει τέλος σε 7 χρόνια ε, πόνου και καταστροφής. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε βεβαίως την Τουρκία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την οποία επισκέφθηκα τον Δεκέμβριο. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν και στην Τουρκία όπου μπορέσαμε να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση επιτόπου, όλες αυτές οι χώρες έχουν ανοίξει τις πόρτες τους ε, στους Σύριους πρόσφυγες με θάρρο παρά τις δικές τους, τα δικά του προβλήματα, τις δικές του προκλήσεις και βασιζόμαστε στην αλληλεγγύη τους απέναντι στους Σύριους πρόσφυγες ε, και βεβαίω και αυτοί βασίζονται στη δική μα αλληλεγγύη από την, την πλευρά της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε. Διότι αυτή, σε, αυτό, σε αυτή την αλληλεγγύη βασίζεται η σχέση μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές άλλες ανθρωπιστικές κρίσεις που ε, αναπτύσσονται στην Αφρική, στην Ιεμένη, όπου έχουμε την πιο έντονη ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή, 22 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος ε, μιας ανίποτης τραγωδίας αθώα θύματα μιας ε, τυφλής ε, μάχης για την εξουσία οι τελευταίες επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύραξη αυτή έχουν δημιουργήσει κάποιες ελπίδες για μια διαδικασία ειρήνευσης εύθραυστη. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε, να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια ακόμα και παρασκηνιακά. Εγώ, η Φεντερίκα, αλλά και ο πρόεδρός μας. Το Μάρτιο θα συμμετάσχω στη διάσκεψη για την Ιεμένη στη Γενέβη, όπου για άλλη μια φορά θα, θα επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας και βεβαίως θα διαθέσουμε ε, και κάποια σημαντικά ποσά χρηματοδότησης Όμω, ε, όπω έχουμε πει από την αρχή, δυστυχώ η ανθρωπιστική κρίση αυτή επιλύεται πολιτικά. Είναι πολιτικές οι λύσεις. Είναι η μόνη απάντηση σε αυτήν την ζωφερή πραγματικότητα. Να μιλήσω τώρα για την Αφρική. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε, αυτό τον, σε αυτή την Ήπειρο η βία και οι φυσικές καταστροφές ε, δημιουργούν ε, ε, καταστροφή και μετατόπιση. Το πιο προφανές παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή του Σαχέλ και οι λίμνες του Τσάντ. Σειράξεις, επιδημίες, κλιματική αλλαγή, κακή διακυβέρνηση, φτώχεια και βεβαίως και η δημογραφική έκρηξη. Πάρα το θέλω αυτό το θέμα, ξέρετε, Ορισμένες φορές θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο σε βάθος για αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας ως ανθρώπου που ασχολούνται με ανθρωπιστικά ζητήματα. Όλες αυτές οι παράμετροι ε, δημιουργούν μια μόνιμα εύθραστη κατάσταση στην περιοχή. Οι ανθρωπιστικές μας προσπάθειες προσπαθούν να καλύψουν ε, τα ζητήματα κακής διατροφής, ε, την έλλειψη τροφίμων, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ζητήματα υγείας για τους πιο ευάλωτους, οι εθνικές κρίσεις ε, μετά στη συνέχεια γίνονται περιφερειακές, αυτό και οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες ανθρωπιστικές ανάγκες, όλο και περισσότεροι μετατοπισμένοι, αναγκαστικά μετατοπισμένοι άνθρωποι, όλο και πιο πολύ ευάλωτοι άνθρωποι απελπισμένοι. Αυτό το έχουμε δει όχι μόνο στην περιοχή του Σαχέλ, αλλά και αλλού και σε άλλες χώρες. Τα τελευταία το τελευταίο έτος είδαμε κάποιες χώρες που αποσταθεροποιήθηκαν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου 60% του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική συνδρομή. Όμως η ανθρωπιστική συνδρομή από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα αισθήματα αυτά. Η Αφρική χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και βιώσιμες λύσεις. Επιτρέψτε μου τώρα να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε κάπως αντισυμβατικά. Πρέπει να δούμε την Αφρική διαφορετικά, όχι όπως συνήθως, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ των ανθρωπιστικ... του ανθρωπιστικού μας και αναπτυξιακού μας έργου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Αφρική. Υπάρχει ένα δικό μας σχέδιο. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τις επενδύσεις ε, εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα μεταξύ άλλων. Πρέπει βεβαίω να είμαστε μετριοπαθείς εδώ, διότι είναι πολλή προσπάθεια ακόμα που μας περιμένει. Να είμαστε μετριόφρονες μάλλον. Και εδώ, επαναλαμβάνω, πρέπει να σκεφτούμε αντισυμβατικά. Τον περασμένο Μάρτι επισκέφθηκα το νοσοκομείο του Μαντζή στο, του Πάντζη μάλλον στο Κονγκό που έχει χρηματοδοτήσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον αγαπητό φίλο του τον Δόκτωρ Μουκουέγγε το βραβείο Νόμπελ του 2018 ένας ε, ε, εξαιρετικός άνθρωπος μεγάλο έργο στον ανθρωπιστικό τομέα τότε οι αρχές δεν, δεν ήθελαν να συνεργαστούν σε αυτό το πλαίσιο Συνδιοργάνωσα τον περασμένο Μάρτιο μαζί με την Ηνωμένα Έθνη και την κυβέρνηση τη Ολλανδία στην πρώτη διάσκεψη για τη δημοκρατία του Κονγκό. Χρηματοδότηση, έτσι. Μπορέσαμε ε, τότε να συγκεντρώσουμε πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή και αυτό ήταν μια τεράστια ανακούφιση για του πιο ευάλωτου ανθρώπου στη χώρα αυτή. Αλλά εδώ είμαστε μεταξύ μα εδώ, στην οικογένεια συζητώ. Πολλέ φορέ ως ε, Επίτροπος για ανθρωπιστικά ζητήματα, ως Ευρωπαίος Επίτροπος και ενώ η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, ένιωσα, μοναξιά σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, τον περασμένο μήνα επισκέφθηκα την Αιθιοπία, μια χώρα που βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ε, υπάρχει ένας νέος πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ξεκινήσει ε, θαραλέες μεταρρυθμίσεις. Στη συνεδρίασή μας ε, εξέφρασα την υπο... υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειές τους για περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία για τους Αιθίωπες. Υπάρχει η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τη γειτονική Ερυθρέα που δημιουργεί νέες ελπίδες για σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή, όμως είναι τεράστιες προκλήσεις ακόμα. 2,7 εκατομμύρια Αιθίωπες έχουν, είναι μετατοπισμένοι, εσωτερικά μετατοπισμένοι λόγω εθνικών σειράξεων. Υπάρχει θέμα κλιματική αλλαγή όλο και περισσότεροι πρόσφυγες που προέρχονται από την γειτονική Ερυθρέα και από άλλε χώρε. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι να υποστηρίξει την Αιθιοπία σε αυτή την κρίσιμη χρονικά στιγμή, διότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα, ένα μοντέλο. Να είναι ένα μοντέλο η Αιθιοπία, ένα παράδειγμα προς μίμηση για και οι άλλε χώρε τη Αφρική. Επίση, επικεντρώσαμε τι προσπάθειέ μα στο Νότιο Σουδάν ε, για φέτο. Μιλάνε από μόνα του, νομίζω, τα δεδομένα, τα γεγονότα. Ανθρωπιστικό χάο σε αυτή τη χώρα απόλυτη απουσία λογοδοσίας των εμπλεκομένων στη σύραξη. Πραγματικά είναι μια ντροπή. Το είπα από την αρχή της θητείας μου. Κάποιοι από τους συνάδελφους εδώ ε, επισκέφθηκαν τη χώρα αυτή. Είναι πραγματικά ντροπή για τη διεθνή κοινότητα. Δυστυχώς οι δύο ηγέτες είναι εντελώς ανεξέλεγκτοι των ε, εμπλεκόμενων πλευρών. Και βεβαίω αυτή η σύραξη απειλεί και τι γειτονικέ χώρε. Την Ουγγάντα, το Σουδάν, Αιθιοπία, Κένια. Ε, είναι μια πρόκληση, είναι μια αμφισβήτηση των δομών του, τη σταθερότητά του. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω καλεί και τι δύο πλευρέ να ξεκινήσουν μια διαδικασία ειρηνευτική για μια συμφωνία για να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφή. Αλλά για την ώρα δεν συμβαίνει κάτι προ την κατεύθυνση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί από εσά ε, επισκέφθηκαν το Cox's Bazaar πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες ε, ζουν εκεί. Επισκέφθηκα ε, την, την περιοχή της Μιαμάρ, το Ράκνιν, την επαρχία του Ράκνιν, λίγο πριν τη μαζική έξοδο. Ε, το επισκέφθηκα εγώ λίγο μετά. τα Ηνωμένα Έθνη μίλησαν πραγματικά για γενοκτονία σε ό,τι αφορά τους Ροίγκα και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, το είδα και με τα μάτια μου. Ε, χαίρομαι που μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επικεφαλή τη προσπάθεια βοηθείας ε, προ Ροχίνγκια και στη Μιαμάρ και στο Μπαγκλαντές και από κοινού με την ΕΕ θα οργανώσουμε μια διάσκεψη για χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση των τον Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει πάνω από 110 εκατομμύρια ω βοήθεια. Στη Λατινική Αμερική τώρα, στη Βενεζουέλα και στα σύνορα μεταξύ Κολομβία και Βενεζουέλα που επισκέφθηκα επίση τον περασμένο Μάρτι, το είδα από πρώτο χέρι, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε την κρίση στη Βενεζουέλα. Τα εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια φέτο. Οι μετατοπισμένοι εντό τη Βενεζουέλα ε, προς γειτονικέ χώρες, ε, ε, οι κοινότητε που τις υποδέχονται. Το Δεκέμβριο ανακοίνωσα μια ενίσχυση 20 εκατομμυρίων ευρώ ακόμα για την ανθρωπιστική κρίση εκεί και γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι της ΕΚΟ κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τη χώρα αυτή και παρασκηνιακά. Τέλος, θέλω να πω δύο λόγια και για την Ελλάδα. Βεβαίω η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα ε, επομίστηκε δυσανάλογο βάρος ό,τι αφορά την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε στο πλευρό του, του ευρωπαϊκού λαού, των ευρωπαϊκών αρχών. Για πρώτη φορά υπήρξε ανθρωπιστική χρηματοδότηση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μέσου ευρω... επίγουσα υποστήριξη με ε, προγράμματα φιλόδοξα, στέγασης, ε, ενίσχυση σε μετρητά όπως το εστία. Παρ' όλα αυτά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, επιτόπου ιδιαίτερα στα νησιά τη Λέσβου και τη Σάμου. Ξέρετε ότι τα ανθρωπιστικά μας προγράμματα στην Ελλάδα θα συνεχιστούν από τις ελληνικές αρχές και από άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν, την DG Home. Αυτό συμφωνήσαμε άλλωστε όταν θεσπίσαμε αυτά τα νέα μέσα και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ε, σε αυτές τις ναπομείνωσες προκλήσεις. ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που υπάρχουν. Θέλω να πω και άλλη μια φορά ότι η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Και βεβαίως ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και πραγματικά πιστεύω ότι η υποστήριξή σας ε, θα είναι κρίσιμη και σε αυτή τη νέα φάση τη ευρωπαϊκή υποστηρίξη προ την Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι, ο αριθμός των σειράξεων ανά τον κόσμο αυξάνονται σε αριθμό, ε, σε διάρκεια και σε περιπλοκότητα. Έτσι λοιπόν η καθημερινή δουλειά τη ανθρωπιστική ενίσχυση είναι όλο και πιο περίπλοκη, όλο και πιο δύσκολη. Η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική έκρηξη επαναπροσδιορίζουν τι ανθρωπιστικέ προσπάθειε τι σημερινέ, ιδιαίτερα στην Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι νέε προκλήσει και γι' αυτό προτείνουμε μια αύξηση 30% στον προπολογισμό, των ανθρωπιστικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. 1,6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όμω όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι τα χρήματα από μόνα του δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε και νέε ιδέε, καινοτόμε λύσει, καλύτερε εταιρικέ σχέσει, συμπράξει και να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά με καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε για να φτάσουμε ε, σε καλύτερες σε μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ ανθρωπιστική βοήθεια, διαχείριση κρίση και πολιτική προστασία. Αυτό είναι και το λογικό και γι' αυτό το RESC EU είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Το RESC EU θα βελτιώσει την απάντηση σε επίγουσε καταστάσει στο εσωτερικό και θα ενισχύσει και την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Έτσι ώστε η ελληνική μα να είναι πιο συνεπή και πιο αξιόπιστη. Με αύξηση του προπολογισμού 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, μικρή αύξηση σε σχέση με τα ωφέλη που θα προκύψουν. Το ανθρωπιστικό τοπίο αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται κάπως ε, προβληματικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις που δεν έχουν προηγούμενο, αλλά κυρίως να ξοδέψουμε καλύτερα τα χρήματα αυτά. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας για το 2019. Όπως πάντα είμαι διατεθειμένος να ακούσω τις ιδέες σας για το πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους από κοινού. Αγαπητή Λίντα, επέτρεψέ μου να πω και δύο λόγια για κάποιους συναδέλφους. Δεν είναι η τελευταία φορά βέβαια που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή Ντεβε, όμως είναι μάλλον ο τελευταίος διάλογος για τις ανθρωπιστικές προτεραιότητες Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια για δύο-τρεις πυλώνες της Επιτροπής σας για τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Λίντα, αξιότιμη πρόεδρε, ο Ενρίκε, ο εισηγητής για, την ανθρωπιστική ενίσχυση και ο Τσαργκέζ που ήταν συντονιστής για τα ζητήματα του έμπολα. Εσύ πάντα με τριόφρον βέβαια, Λίντα, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είχες μια πολύ δίκαιη αντιμετώπιση μεταξύ πολιτικών, μεταξύ συναδέλφων. Ε, είχες όραμα, ενέργεια και δέσμευση στην Προεδρία σου. Ήσουν ένα σύμμαχος κλειδί για να μπορέσουμε να κινηθούμε γρήγορα, να διαθέσουμε τα χρήματα αυτά. Εργάστηκες άοκνα για την κινητοποίηση χρημάτων, χρηματοδότησης απέναντι σε πολλές κρίσεις που δεν είναι πια στα προσελίδα των εφημερίδων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η Λίντα πραγματικά έφερε στην ε, πρώτη γραμμή την ανάγκη καλύτερων λύσεων, πιο μακροπρόθεσμων σχεδιασμών και βεβαίως ήταν στο πλευρό μας όταν η Ελλάδα είχε κατακλειστεί από πρόσφυγες ε, για να δημιουργηθεί ιδιαίτερα αυτό το εργαλείο επίγουσας στήριξης. Ευχαριστώ Λίντα γι' αυτό. Να, να και στη συνεισφορά σου στις συζητήσεις για το Global Compact ε, των ΗΕ Εθνών ε, για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, τη βία, ενώ υπήρχε αρκετά μεγάλη επιφυλακτικότητα ακόμα και από τα κράτη-μέλη μας από την, πλευρά, από την αρχή της θητείας μου κατάλαβα ότι μπορούσα να βασιστώ σε σένα όχι μόνο ως συνάδελφος αλλά και ως αξιόπιστος και πιστός φίλος και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Φίλε μου Ενρίκια ένας πραγματικός υπερασπιστής των ανθρωπιστικών μας αρχών, ένας σύμμαχος ε, στο θέμα της εκπαίδευσης σε επίκους καταστάσεις, πάντα ψάχνοντας τις καλύτερες ε, λύσεις ε, για την ε, ε, καλύτερη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικού και ανεξιακού τομέα. και θυμάμαι την κοινή μας δράση στην ανθρωπιστική σύνοδο στην Σανγκάη, στην Κανκούν και στην Κωνσταντινούπολη. Πάντα ήσουν ένας αξιόπιστος εταίρος για να, βρεθούν, να βρεθεί χρηματοδότηση για, για την απάντηση σε κρίσεις. Με τον ισπανικό δυναμισμό σου πάντα είχες αυτή την παραπάνω ενέργεια ε, που βοηθούσε στις κρίσιμες στιγμές. Και οι δυο σας ε, πραγματικά ε, πιστέψατε στο διάλογο, στη συμμετοχή. Θα μου λείψετε διότι έχετε υπερασπιστεί τις ανθρωπιστικές αξίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επίσης ε, να εκφράσω τις ειλικρινές μου ευχαριστίες και στους δυο σας αλλά και σε όλους τους συναδελφούς που είναι εδώ σήμερα και όπως πάντα είναι τιμή και χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί σας παρά το λέω αυτό δεν είμαι καινούριο ε, στον πολιτικό κόσμο έχω εμπειρία και ευθύς εξ αρχής ε, στη συνεργασία μας είδα ότι μπορούσα να βασιστώ σε εσά ε, σε πολύ δύσκολε, σε πολύ απαιτητικέ αποστολέ, Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και βεβαίω είμαι εδώ για να συζητήσουμε και αυτό το έτος, του προγραμματισμό αυτού του έφους που δεν είναι δύσκολος για όλους μας. Ναι, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες έτσι κι αλλιώς ε, να μιλήσουμε, αλλά σε ευχαριστώ πραγματικά Χρήστο. Στην πρώτη ακρόαση μείναμε με το στόμα ανοιχτό όταν ε, καταλάβαμε την εμπειρία που είχες για θέματα αυτά και όταν είδαμε μετά και τι συνέβαινε στη χώρα σου και πώς το αντιμετώπισες και όλα αυτά. κατανοεί σε όλα τα προβλήματα με ε, ευαισθησία και ανθρωπισμό. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Ελίκη Γκερέρο, ο οποίος ε, είναι ο εξέχων και έξοχος συντονιστής μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τα φιλικά σας ε, λόγια ε, και τα θετικά λόγια που είπατε ε, για μένα και έτσι δυσκολεύομαι να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω γιατί εγώ ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για την εργασία σας ενώ τώρα θα φανεί λίγο σαν ε, να σας λέω καλά λόγια για να ε, είμαι ευγενής επειδή εσείς μου απευθυνθήκατε με αυτόν τον τρόπο αλλά πραγματικά σας λέω και πριν ακούσω αυτά που είπατε, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αναφερθήκατε στην Επιτροπή μας, που είναι λίγο η οικογένειά σας. Είναι αλήθεια ότι οι οικογένειες είναι περίπλοκα συστήματα και πολύ συχνά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά μεταξύ των μελών ε, ας πούμε όλοι βλέπουν με φρίκι το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό δείπνο όπου μπορεί να ακουστούν ε, φρικτά πράγματα ε, και όπου ξαφνικά μέσα από τη συζήτηση ας πούμε φουντώνει μία λογομαχία. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν αυτή η ίδια οικογένεια έχει σοβαρά προβλήματα ή όταν αντιμετωπίζει δυστυχίες ή προβλήματα, η οικογένεια ενώνεται. Και εμείς σε αυτή την Επιτροπή και όπως και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύουμε ε, με τη δυστυχία χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων ανθρώπων, πραγματικά είμαστε ενωμένοι γιατί ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυστυχίες, αυτές τις περίπλοκες καταστάσεις που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μια επιτροπή πολύ πιο προοδευτική εντό εισαγωγικών ε, από το σύνολο του Κοινοβουλίου, γιατί εμείς δουλεύουμε με ανθρωπιστικά ε, θέματα και είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτά. Αφού τα είπα αυτά, όμως πιστεύω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω για την εργασία που κάνατε ως Επίτροπος και για τη σχέση σας με το Κοινοβούλιο γιατί εγώ συμμετέχω και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, αλλά Ξέρετε, δεν συνηθίζεται ένας επίτροπος να έρχεται τόσο συχνά σε επαφή και να κάνει τόσες συνεδριάσεις με το σύνολο των μελών της Επιτροπής ε, ή ε, να έχει επαφές με μεμονωμένους βουλευτές ε, αυτής της Επιτροπής και όχι μόνο εντός των τυπικών διάβλων. Επιπροσθέτως, ε, κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε πολύ καλά πώς να δράτε επί τόπου, επί του πεδίου δηλαδή. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πραγματικές απαντήσεις μπορεί να βρει κανείς όσον αφορά τις ανθρωπιστικές κρίσεις παρά μόνο επιτόπου και όχι από το γραφείο του ή όχι διαβάζοντας ή γράφοντας ψυχρές στατιστικές. Θα πρέπει κανείς να είναι επιτόπου, θα πρέπει να βλέπει τους ανθρώπους, θα πρέπει να αγγίζει τη δυστυχία που αντιμετωπίζουν από κοντά έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει λύση. Ένα σημαντικό τμήμα της παρέμβασής σας αφορούσε την αναφορά πορών ε, στοιχείων ε, και μαχών που δίνονται είτε για την εκρίζωση του έμπολα, είτε για τη βοήθεια κάποιας χώρας, είτε για την ε, Βενεζουέλα όπου διαπιστώνεται τα προβλήματα ε, άλλες ε, χώρες ε, της μεσημβρινής Αφρικής που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε γιατί υπήρξατε επίτροπος ο οποίος πραγματικά ήταν παρόν στα πεδία της δράσης. Είχαμε επιτυχίες ε, τα τελευταία χρόνια και αναφερθήκατε σε αυτά, ε, εκπαίδευση σε κρίσιμες καταστάσεις. Ας πούμε, καταφέραμε να φτάσουμε στα 55, συγγνώμη, 5,5 εκατομμύρια ε, παιδιών που παρότι βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης καταφέρνουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους γιατί ε, αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι απολύτως απαραίτητο και για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα άμεσα προβλήματα και τις άμεσες ε, κρίσιμες καταστάσεις που έχουν απέναντί τους, αλλά και για να οικοδομήσουν το μέλλον τους. Επίσης, 300 ε, ε, χιλιάδες ε, ε, Σύριοι από την Τουρκία επιστρέφουν σιγά σιγά και αυτό πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που δώσαμε στα πιο μικρά παιδιά δηλαδή την δυνατότητα να εκπαιδευτούν. Αναφερθήκατε στην έμπολα, αναφερθήκατε ε, στην ε, ε, βία κατά των γυναικών, αναφερθήκατε στον έξους, στο κόξ κλπ. Τα ξέρουμε και αυτά. Επίσης ξέρουμε ότι διδαχτήκαμε από τα λάθη μας. Διδαχτήκαμε ότι σημαντική είναι η πρόληψη όταν μιλάμε για μείωση φυσικών κινδύνων. Επίσης, μάθαμε ότι κρίσεις όπως αυτή ε, του έμπολα δεν ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν δεν δημιουργηθούν στις χώρες που χρειάζονται οι απαραίτητες ιατρικές δομές και ε, επίσης ε, υπάρχουν θέματα τα οποία λύνονται μόνο και μέσα πολιτικών, μέσω πολιτικών λύσεων και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει την λύση αυτή. Μάθαμε επίσης ότι υπάρχουν και σημαντικά πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσουμε περισσότερο και από πιο στενά την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπο αυτής επί των ανθρωπιστικών κρίσεων Ξέρουμε ότι μπορεί να έρθει ένα νέο φαινόμενο ελνίνιο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα ε, ε, σε περιοχές μάλιστα που μπορεί να βρίσκονται αρκετά μακριά από αυτές που ε, πλήττονται από το καιρικό φαινόμενο. Επίσης έχουμε το επόμενο MFF που οπωσδήποτε είναι σωστό να έχει και την δυνατότητα να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Επίσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις τοπικές οργανώσεις που πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Γνωρίζουμε και από τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δουλεύουν σε περιοχές δύσκολες ότι ε, χωρίς βοήθεια στις τοπικές οργανώσεις δεν πρόκειται να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ε πιο μεγάλες ε, και τις ντόπιε ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν βλέπουμε τη μεθοδολογία των βοηθειών που μπορεί να δώσουμε και της αρρωγής μας. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε νέες ασθένειες ή την επανεμφάνιση παλαιών ε, και εξαφανισμένων μέχρι τώρα ε, ασθενειών. Γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει επίσης το φαινόμενο της ισχυρής αντίστασης σε ιούς και επομένως Καταλαβαίνετε ότι σε χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, αλλά και σε άλλες πολλές χώρες μπορεί να ξαναβρούμε ασθένειες που πιστεύαμε ότι είχαν εκκριζωθεί. Δύο τελευταία σχόλια. Ένα το οποίο αφορά τις ε, δεσμεύσεις ε, που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κωνσταντινούπολη, στην ε, διάσκεψη κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σαν ένωση, αλλά και δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια στην επόμενη ε, πολιτική περίοδο, στον επόμενο πολιτικό ε, κύκλο, έτσι ώστε ο απολογισμός να είναι θετικός. περαίνουμε κάτι το οποίο ε, ε, ανέφερε και ο κύριος Επίτροπος, Αφρική. Ζω στην Ισπανία και μπορείτε να φανταστείτε ότι για μας ε, η Αφρική πραγματικά είναι το σύνορό μας. Είναι έξω από την πόρτα μας. Δεν θα αναφερθώ στους πρόσφυγες ε, και τους μετανάστες που φτάνουν αυτή τη στιγμή λόγω αλλαγής ε, των ε, οδών στην Ισπανία. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, η Ισπανία είναι ε, μια πλούσια χώρα με πολλά εκατομμύρια κατοίκους. Αλλά εμείς ως ε, χώρα γνωρίζουμε ότι ε, ε, εμείς είμαστε το τελικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Αφρική, ότι γείτονά μας είναι η Αφρική και επομένως θα πρέπει να λύσουμε προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μονάχα με την αναπτυξιακή βοήθεια ή με χρήματα ή με προγράμματα. Μόνο με δικαιοσύνη, μόνο εάν είμαστε δίκαιοι απέναντι στην στην ε, χώρα, στις χώρες αυτές, απέναντι στην Ήπειρο αυτή, εάν ε, ε, πραγματικά ακολουθήσουμε τις συμφωνίες Κοτονού, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλές σχέσεις με την Αφρική. Θέλω να υπενθυμίσω ότι κάποια στιγμή είπατε ότι ως Επίτροπος πολλές φορές αισθανθήκατε μόνος και ελπίζω ότι θα είστε λίγο λιγότερο μόνος μετά από την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ, Ενρίκε, η Χαϊδη Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα της αναγνώρισης και εμείς εκτιμούμε το έργο σας και τη παρουσία σας εδώ για να μας δίνετε αναφορά. Είπατε ότι θα θέλατε κάποια μέρα να μιλήσετε λίγο περισσότερο για τα δημογραφικά... κάποια μιλάνε δημογραφική έκρηξη δεν ξέρω εσείς τι άλλα χρησιμοποιήσατε, αλλά δεν ήθελα να τη χρησιμοποιήσω. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε λέξεις που θυμίζουν βόμβα για τις δημογραφικές τις ε, μέγες εξελίξεις περιοχές που περιγράψετε. Απλά θα ήθελα να ακούσω τι τις απόψεις σας, γιατί έχετε δει πολλά πράγματα επί που έχετε ακούσει πάρα πολλές ιδέες σίγουρα για το τι πρέπει να γίνει. Τι συμβουλές έχετε να μας δώσετε λοιπόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Ένα σημείο είχα εγώ Μάλλον το ένα ήταν αυτό που είπαν Ρή και για τον ρόλο των τοπικών ΜΚΟ σε καταστάσεις ε, έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει σχετική έκθεση που, που να είναι, θα δημοσιοποιηθεί, αλλά σίγουρα οι ΜΚΟ πολλές φορές εργάζονται υπό πολύ δυσχερείς συνθήκες ε, και οι άνθρωποι εκεί ε, μπορούν να δώσουν τη βοήθεια στις τοπικές κοινωνίες. Για τη Συρία, για παράδειγμα, το να τους στείλουμε εκεί είναι δύσκολο να στείλει κανείς ε, εργαζομένους ε, που εργάζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό και για την Ελλάδα είναι το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, στηρίξατε την Επιτροπή μας και εμείς σας υποστηρίξαμε στην ιδέα σας να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα. Όταν ήταν ε, πολύ ψηλές οι αφήξεις προσφύγων από τη Συρία. Ακούμε όμως κάποια πολύ ανησυχητικά ε, πράγματα για την κατάσταση των προσφύγων στη Λέσβο και τη Σάμου. Ιδίω σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές το έχουμε θέσει και στα Υπουργεία, τα ελληνικά. Αλλά και στα τέλη Δεκεμβρίου, ε, οι που παίρναμε είναι ότι τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Αντιθέτως, έχω μιλήσει με τον Επιτροπό Αβραμόπουλο και έχω ζητήσει και τον πρόεδρο τη Επιτροπή Λίπε τον Κλοντ Μωρέ, να το βάλει στη μέση διάταξη όταν θα έρθει πρώτο για να τα συζητήσουμε και μαζί του. Διότι εμεί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και το σωστό είναι να ε, κάνουμε τα σωστά. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά. Πρέπει να του δοθεί ιδέουσα προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τι ελληνικέ αρχέ. Γνωρίζουμε τι δυσκολίε. Εγώ έχω μεταβεί στη Λέσβο μου είπανε ότι κάθε μέρα φτάνουν 35.000, ε, κάποιες εβδομάδες ήταν αυτά τα νούμερα καθημερινά. Ε, η δουλειά που γίνεται είναι τρομερή, σίγουρα. Τώρα όμως έχουν πέσει πολύ τα νούμερα και θα πρέπει ο κόσμος εκεί να έχει τις σωστές συνθήκες διαβίωσης. Ελπίζω αυτό να γίνει και ελπίζω και εσείς να συνεχίσετε να πιέζετε και εμείς να συνεχίσουμε να ε, ρωτούμε το Παρακαλώ, έχετε το λόγο, Επίτροπε, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ευγενικά σας λόγια. Γνωρίζετε. Και το είπα. Όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ένιωθα ότι με υποστηρίζετε υπό την ιδιότητά μου και ακόμη και όταν βρισκόμουν επί τόπου και για μένα αυτό ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτή η βοήθεια. Ήταν σημαντική ιδίω στι αποστολέ που είχαν αντιμετωπίσει δυσκολίε όπω ότι ο Σουδάν για παράδειγμα και στο Κονγκό ή την Ιγυρία εκεί που έχουμε τη δράση της Μποκοχαράμ ήξερα την υποστήριξη που έχω από εσά ως συνάδελφου και ως βουλευτέ με υποστηρίζετε και αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Γιατί έτσι μπορούσα να τα πω έξω από τα δόντια για τα προβλήματα επιτόπου. Και κάτι τελευταίο για τις σχέσεις μας. Ε, ναι, θα προσπαθήσω να το ξανακάνω, να το τονίσω εκ νέου αυτό. Ξεκινώ από την ερώτηση της Λίντα για την Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψω τώρα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Γιατί θέλω πολλά να πω. Γνωρίζω πολύ καλά άλλωστε την κατάσταση επιτόπου. Η κατάσταση ειδικά στη Λέσβο και στη Σάμο ε, δυστυχώς παραμένει προβληματική. Όπως ε, και η Λίντα ήδη είπε, οι ελληνικές αρχές, οι τοπικές αρχές, ο πληθυσμός έκανε μεγάλες προσπάθειες. Και ειλικρινά την τελευταία εβδομάδα είδαμε και τον θάνατο αυτό της εξαιρετικής γιαγιάς η οποία περίμενε τα προσφυγόπουλα για να τα βοηθήσει να πιούν λίγο γάλα και να επιβιώσουν. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είδαμε και στι συναντήσεις μου με τους ε, κατά καιρού υπουργούς για τη μετανάστευση ε, προσπάθησα πάρα πολύ έτσι ώστε να μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην υπηρετική Ελλάδα γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η λύση θα δοθεί μέσω του προγράμματος που εγκαθιδρύσαμε του εστία, του λεγόμενου εστία. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν τρία σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αυτού του θέματος. Το πρώτο υπάρχει ένα φατίκ ε, από τις τοπικές κοινωνίες και είναι αναμενόμενο. Το δεύτερο είναι ότι η συμφωνία, το EU Turkey Facility, περιλαμβάνει αυτή την διατύπωση ότι μπορούν να επιστραφούν πίσω πρόσφυγες στην Τουρκία οι οποίοι βρίσκονται στα Aegean Islands, στα νησιά του Αιγαίου. Και αυτό είναι μια συνθήκη η οποία περιορίζει τις επιλογές. Το τρίτο σημείο που θέλω να δείξω που είναι θετικό κατά την άποψή μου είναι ότι όσες φορές μπορέσαμε να μεταφέρουμε οι ελληνικές αρχές να μεταφερθούν πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα ε, και ήταν Σύριοι πρόσφυγες γιατί υπάρχει άμεσα ή έμμεσα μία διάκριση μεταξύ Σύρων προσφύγων και των υπολείπων Αφγανών και άλλων, ε, υπήρξε όντως παραδειγματική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων και εντάχθηκαν όλοι σε δομές φιλοξενίας οι οποίες ήταν, ήταν πολύ καλές. Που σημαίνει, επειδή τα δικά μου σερβίσε στην DG θα φύγουμε με βάση το πρόγραμμα του, του instrument, Μάρτι-Απρίλη. Είμαι σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την DigiHome για να μπορέσουμε και τι ελληνικές αρχές αυτή η περίοδος συμμεταβατική transit period να είναι όντως πολύ αποδοτική και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όσο πιο πολλούς πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία με την DigiHome Home για να κάνουμε πολλά προγράμματα που αφορούν στα παιδιά, τις single mothers και ε, ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης. Καταληκτικά θα έλεγα ότι στην Ελλάδα παρόλη την προβληματική εικόνα έχουν επιτευχθεί περισσότερα από όσο αποτυπώθηκαν είτε μέσα από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ είτε μέσα από πραγματική παράθεση στοιχείων. Έτσι είναι πολλές φορές η σκληρή πραγματικότητα που τα καλά μια κοινή προσπάθειας δεν παρουσιάζονται και παρουσιάζονται τα, καλά, τα κακά που υπάρχουν. Αλλά θέλω να είμαι τίμιος και ειλικρινής με τις ελληνικές αρχές. Έκαναν όντως μεγάλες προσπάθειες. Αλλά υπάρχουν και παραμένουν πολλές ακόμα αδυναμίες ανεξάρτητα εάν η DG ECO αποχωρήσει από την Ελλάδα τους επόμενους μήνες, προσωπικά παραμένω δεσμευμένος να συνεχίσω τις επαφές μου με τις ελληνικές αρχές εξαιτίας και της ελληνικής μου ιδιότητας ως Κύπριος Έλληνας για να βοηθήσω όσον μπορώ έστω και στο παρασκήνιο όπως λέμε, behind the scene, για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να καλυτερεύσουμε την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. I would like to... Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για την παρέμβαση του Ενρίκη και ιδίως σε σχέση με τις τοπίες ΜΚΟ και τους ε, ντόπιου ε, εργαζόμενους ε, στο πλαίσιο ανθρωπιστική βοήθειας. Το ανέφερε και η Λίντα και συμφωνώ μαζί σου Λίντα ότι χωρί τη δική τους υποστήριξη και τη δική τους ε, προσήλωση και αφοσίωση είμαι βέβαιο πως το ανθρωπιστικό έργο εμείς που επιτελούμε επί σε πολλές χώρες που δέχονται ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Διότι γνωρίζουν αυτοί καλύτερα από σε εμάς τις δυσκολίες. Το είδα ε, στην Ιορδανία, στην Μπεκά, ε, στο Ιράκ, έξω από τη Μοσούλη, το είδα και στην Τουρκία, φυσικά βέβαια και στην Αφρική. Επομένως, πρέπει να εξεύρουμε τρόπους ε, ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Και βέβαια είμαστε ενώπιον διλήμματος. Πρέπει να τηρήσουμε τους δικούς μας κανόνες, και κανονισμούς με βάση συμβουλέ ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα να εξεύρουμε και τρόπους ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να αξιοποιήσουμε πιο συγκεκριμένα ε, με πιο συγκεκριμένο τρόπο τις τοπικές ΜΚΟ. Οι διεθνείς ε, οργανισμοί, οι οργανισμοί του ΟΗΕ, οι διεθνοί μας δηλαδή, συμφωνούν απόλυτα με την προσέγγιση αυτή. Με την δική σας υποστήριξη λοιπόν Μεταξύ άλλων νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πιο ευέλικτους τρόπους, ώστε όλο και περισσότερο να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια τοπικές ΜΚΟ. Αυτό είναι για μένα προϋπόθεση, αν θέλουμε η ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου να είναι αποτελεσματική. Ταυτόχρονα βέβαια, το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Ενρίκε, γιατί με τις ΜΚΟ, τις τοπικές, μειώνεται και το πάγιο κόστος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανθρωπιστική κοινότητα. Διότι πρέπει να δεχθούμε το ότι δεχόμεθα επίθεση από λαϊκιστές και λοιπούς που δυστυχώς επιμένουν πως η ανθρωπινιστική και η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα είδος πολυτέλειας για τους Ευρωπαίους και στην προεκλογική στρατηγική της τις πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα όλοι μας και να αγωνιστούμε σε αυτές τις ευρωεκλογέ και την προεκλογική εκστρατεία για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με τη στάση αυτή απέναντι στην ανθρωπιστική αναπτυξιακή βοήθεια. Αφρική, συμφωνώ απόλυτα. Θα ήθελα ωστόσο να πω δύο λόγια παραπάνω για την πραγματική ανησυχία που έχω σε ό,τι αφορά την πληθυσμική έκρηξη. Όπως είπα, Είμαι πεπισμένος πως η μεγαλύτερη πρόκληση για όλους μας είναι η Αφρική, ιδίως για την Ευρώπη βέβαια. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται μια παγκόσμια αντίδραση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά είναι παγκόσμιο, άρα πρέπει να σκεφτούμε, όπως είπα, αντισυμβατικά και όχι με μια προσέγγιση business as usual. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, η προσέγγιση μας πρέπει να περιλαμβάνει την παραδοχή του ότι οι αφρικανικές χώρες είναι εταίροι και πρέπει κάπως αυτή τη μεταπικιακή ε, προσέγγιση η τη φιλανθρωπική αγαθοργή προσέγγιση να την ξεπεράσουμε. Δηλαδή πρέπει τους Αφρικανούς ε, ηγέτες Αφρικανικής Αφρικανική να τους δούμε ως και να συζητούμε μαζί τους πολιτικά για την διακυβέρνηση ή τη μη διακυβέρνηση καλύτερα για τη διαφθόρα και τη δημογραφική την πληθυσμιακή έκρηξη. Αυτό το ερώτημα, το θέμα το έχω θέσει σε ορισμένου ηγέτε και για να είμαι ειλικρινή, ήταν πολύ θετική η απήχηση που συνάντησε και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, το γνωρίζω από την δική μου χώρα, πως ο γενικός προγραμματισμός σε ό,τι αφορά την πληθυσμική έκρηξη, δεν είναι αντίθετο με τα ε, ηθικά, με, με τι ηθικέ μα αρχέ και το ηθικό μα πλαίσιο. Εγώ δεν έκανα ποτέ ε, μία πρόταση κάτι που να μοιάζει με την κινέζικη προσέγγιση, ε, μακριά από μένα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους και μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε καλύτερους τρόπους για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ίσως δε είμαι βέβαια στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, ανθρωπιστική βοήθεια αφορά πιο πολύ την αναπτυξιακή βοήθεια και τις επενδύσεις μας προς την Αφρική. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε την αναπτυξιακή μα βοήθεια να την συσχετίσουμε με συγκεκριμένα κριτήρια για την μη και διακυβέρνηση και την διαφθορά. Ταυτόχρονα. Φυσικά και πρέπει να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. από πείρας προσωπικής, καθότι κατάγομαι από την Κύπρο, που είναι ένα σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο, μπορώ να σας πω πως το μοντέλο των ΣΔΙΤΑ, των συμπράξεων δημόσιο ιδιωτικού τομέα, είναι πολύ αποτελεσματικό μοντέλο για να συμμετέχει ο ευρωπαϊκός ιδιωτικός τομέας και για να γίνει αυτή η προσπάθεια αντιμετώπιση ε, της μη διακυβέρνηση ε, και της διαφθοράς. Πρέπει να τα πούμε αυτά στου αφρικανού εταίρου μας, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Τα συζήτησα με τον νέο Αιθίωπα Πρωθυπουργό. Είναι ένας νέος ηγέτης που είδα ότι είναι πραγματικά έτοιμος να δεχθεί νέες ιδέες και να δει μια διαφορετική εταιρική σχέση με εμά. Και στην πρώτη μου παρέμβαση εστίασα στο ότι ίσω δούμε ένα είδο αιθιοπικού μοντέλου για την Αφρική συνολικά. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. a big, um, a big Ευχαριστούμε πολύ κύριε που Μας καλύψατε ε, όλη την Ήπειρο ουσιαστικά, ε, μάλλον όλο τον πλανήτη και δείξατε πόσο σας συναρπάζουν τα θέματα αυτά για τη δημογραφική εξέλιξη. Ξέρετε ότι δεν έχουμε και τόσες επιλογές οι γυναίκες, ε, μειώνονται ε, οι επιλογές. Θα δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες, ε, που, οι αριθμοί μάλλον, που οι γυναίκες δεν έχουν τις επιλογές. Βλέπουμε. Επίτροπος. Πάντα εστιάζω στην εκπαίδευση σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Είναι εκπαίδευση σημαντική και στον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω. Θα σας ξαναδούμε σίγουρα ε,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 για την ερώτησή σας. Η απάντηση είναι ότι η ΔΑΚ ε, έχει ξεκινήσει την, τον εξυγχρονισμό ε, της μεθοδολογίας το 2012 και τα αποτελέσματα είναι καλά. Το 2014 σε μια συνεδρία υψηλού επίπεδου η ΔΑΚ ε, αναγνώρισε ότι υπάρχουν νέες τάσεις στην βοήθεια και την ανάπτυξη. Αποφάσισε να υπογραμμίσει περισσότερο το ρόλο των ίδιων πόρων καθώς επίσης και τις εγγύσεις που θα πρέπει να δίνονται ε, στον τομέα της, ε, των ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων. Και στην μπεμπα. αυτό επιβεβαιώθηκε στα πλαίσια και του θεματολογίου του 2030 και του στόχους όπου με αυτό συνδέονται αξιολογείται η υψηλή ε, σημασία των ε, δανείων καθώς επίσης ε, και οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Η ποσοτική μέθοδος εφαρμόζεται το 2019 για το reporting του 2018. Ε, σχέδια διεύρυνσης αυτών των ε, μεθόδων και προς τον ε, ιδιωτικό τομέα δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες οργανωτικής διαφοροποίησης. Θεωρεί ότι ο εξυγχρονισμός των ε, της μέτρησης των στόχων ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τα εργαλεία του ιδιωτικού τομέα, ε, όπως αναφέρεται και σε την επιστολή που περιλαμβάνεται στην ερώτηση, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, κοιτάξουμε από πολύ κοντά τις συγκεκριμένες μορφές συναλλαγών που μπορεί να είναι πιο προβληματικές. Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε η προσθετικότητα να εφαρμόζεται μονάχα όταν υπάρχει η ρήξη της αγοράς ή η ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων. Ο κίνδυνος ε, το, της αναφοράς μη συνενετικών ε, πράξεων αναφέρεται επίσης. Η Κομισιόν προσπαθεί να βρει ε, συμβιβαστικές ε, λύσεις ε, μεταξύ των μελών ΝΤΑΚ και της άλλης πλευράς. Υπάρχει μια ενδιάμεση λύση, μια και ελήψη τελικής συνολικής λύσεως, η οποία βασίζεται στην, στο cash flow, στην ροή. Συνεχίζεται η ανάλυση. Ε, και από την γραμματεία. Αυτή τη στιγμή ε, ε, και για τα δάνεια σε grant equivalent αλλά και στον έλεγχο cash flow είναι μια συμβιβαστική λύση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Χάιντι Χαουτάλα. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέει η Κομισιόν είναι ότι ε, έγινε κάποιο λάθος ε, από τους προηγούμενους προέδρους της ΝΤΑΚ σε σχέση με αυτό που αναφέρεται στην επιστολή. Όντως είναι έτσι. Επίσης, θα μπορούσατε να πείτε ότι τα εχέγγυα έχουν, ε, που έχουν ληφθεί στα πλαίσια του συμβιβασμού είχαν σαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει ενιαία ε, μορφή και ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, απομακρύνονται από την έννοια της conditionality συγκεκριμένων προϋποθέσεων δηλαδή και πηγαίνουν προς την additionality, στην προσθετικότητα. Πολύ σύντομα να απαντήσετε αν είναι δυνατόν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Ναι, Πράγματι θεωρούμε ότι η ανοιχτή επιστολή δεν ε, είναι σωστή και όντως έχουν ληφθεί υπόψη τα εχένια. Μπορεί ε, να υπάρχει αυτή η συμφωνία, ε, υπάρχει αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί για το cash flow, η οποία θα εφαρμοστεί για τον ιδιωτικό τομέα και στην ενδιάμεση περίοδο όλα τα κράτη-μέλη ήταν υπέρ ε, και της additionality και της ε, concessionality και αυτό δεν ήταν πρόβλημα, το πρόβλημα ήταν αλλού. Ε, στο λεγόμενο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο discount rate, το οποίο πρέπει να υπολογιστεί με συγκεκριμένο τρόπο. Η Γερμανία και η Γαλλία ιδιαίτερος ζητούσαν υψηλότερα ποσοστά. Η Ισπανία ε, ζητούσε χαμηλότερα ποσοστά και δεν βρέθηκε συμφωνία εντός της ΔΑΚ. Επίσης ε, ε, και άλλες μη ενωσιακές χώρες είχαν διστάμενες απόψεις όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Εντάξει, δυστυχώς ε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ε, ε θέλεις, και μια, ε, θέλεις και γραπτά την απάντηση. Ωραία, παρακαλώ να μας στείλετε λοιπόν αντίγραφο της απάντησής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα διάφορα δεν έχουμε κάτι. 25 η επόμενη συνεδρίαση. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα μία για την Ιεμένη, μετά άλλη μία για την, ε, με το ηλεκτρικό συνέδριο. Α, ναι, όχι, έχουμε 7 Φεβρουαρίου την επόμενη συνεδρία σήμερα, Θα σας τα στείλουμε και γραπτά αυτά. Δεν χρειάζεται να τα πούμε από τώρα. Και Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτήν την συνεδρίαση και θα πάμε σε μια συνεδρίαση άλλη από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην αίθουσα 2Q2. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκεί θα μιλήσουμε για ε, τη θέσπιση του νέου μηχανισμού.